Η κυρία Κόστιγκερ μου είπε ότι πρέπει επιτέλου να ξεκινήσουμε. Και τη είπα εντάξει. Decision is important for us. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προεόρτη εβδομάδα για μας. Αλλά ακριβώ ε, το γεγονός ότι ακολουθούν διακοπές θα επιδράσει θετικά και τις εργασίες μας. Το πρώτο σημείο είναι η έγκριση μέρης της διάταξης. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Όχι. Ανακοινώσεις. Έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσε, με εξαίρεση τα τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και εγωεδελικά. Αναμεταδίδεται και απευθεία στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Μάλιστα, η έγκριση των πρακτικών τη 13 η Φεβρουαρίου θα γίνει με την συνήθη διαδικασία. Περνάμε στο σημείο 4, το πρώτο κύριο θέμα, πρώτο ουσιαστικό μάλλον θέμα τη απογευματινή συνεδρίαση, που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Bernhard Ούρλα εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας των Τροφίμων, του ΕΦΣΑ. Αυτό αποφάσισαν οι συντονιστές, να καλέσουμε τον εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων, για ανταλλαγή απόψεων για να δούμε τις εργασίες αυτού του σημαντικού οργανισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επαναλαμβάνω, ο οργανισμός αυτός είναι πολύ σημαντικός, ε, ιδιαίτερα για τη συμμόρφωση με το δίκαιο που διέπει την ασφάλεια των τροφίμων. Και μάλιστα εκπονεί σημαντικές επιστημονικές μελέτες ε, για τις απειλές στην επιστηστική ασφάλεια, έχει εμπειρογνώμονες για την ποιότητα τροφίμων και γενικώ ε, έχει ως αρμοδιότητα το πολύ αυτό σημαντικό θέμα της ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλύει τον επιστημονικό κίνδυνο, τον διαχειριστικό κίνδυνο, την πολιτική δηλαδή, γιατί η αξιολόγηση κίνδυνο γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο. Οπότε είναι πολύ σημαντικές οι αρμοδιότητες του οργανισμού αυτού και δεν αξιοποιούμε στο έπακρο τη δυνατότητα συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Αυτοοργανισμό. Αλλά δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον δόκτωρα Ούρλ που θα μας παρουσιάσει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες του οργανισμού ΕΦΣΑ θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Κύριε Διευθυντά, είμαστε όλοι αυτιά. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω το λόγο επισήμως σαν εκτελεστικός διευθυντής της ΕΦΣΑ εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας και να θα ακολουθήσει και ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν πολλές επικαλύψεις μεταξύ αυτού που κάνουμε και της Επιτροπής σας. Αυτά που κάνετε είναι πολύ χρήσιμα για μας και ασχολούμαστε με την ευημερία των ζώων, με θέματα φυτοπροστασίας, τροφίμων και φυσικά αυτό ο ανήκει στην δική μας αποστολή καθώς και η αξιολόγηση και η εκτίμηση των κινδύνων. Θα ξεκινήσω με κάποια εισαγωγικά σχόλια. Θα μιλήσω πρώτα απ' όλα για τις δραστηριότητές μας που μπορεί να στηρίξουν και τη δική σας εργασία. Θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα και κατόπιν θα μιλήσω λίγο για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της επιστήμης, της πολιτικής, πώς προετοιμάζουμε τις επιστημονικές μας γνωμοδοτήσεις και πώς αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αποφάσεων και την ομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, εδώ θα πρέπει να σας πω ότι μετά από την κρίση της σποκώδης εγκεφαλοπάθειας ιδρύθηκε ο οργανισμός μας, ο ΕΦΣΑ ο καθότι θέλαμε να ξεχωρίσουμε την αξιολόγηση του κινδύνου από τη διαχείριση των κρίσεων. Η αξιολόγηση των ε, κινδύνων για την ε, ασφάλεια των ειδών διατροφής έπρεπε να είναι κάτι διαφορετικό από τη διαχείριση της κρίσης. Πρόκειται για μια επιστημονική εργασία που αφορά την τροφική αλυσίδα και πρόκειται για κάτι που έχει σχέση με την εμπιστοσύνη. Διότι αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην τροφική αλυσίδα, στα τρόφιμα, κινδυνεύουμε να μην μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά και τις κρίσεις. Ήταν για μας λοιπόν πολύ σημαντικό να ελέξουμε το θέμα των διαδικασιών, των δεδομένων και βεβαίως να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που συμβαίνουν στι Ηνωμένε Πολιτείες, στον αντίστοιχο οργανισμό, στην FDA. Είναι κάτι που θα έλεγα συμβαίνει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εμείς θελήσαμε να δημιουργήσουμε με 450 άτομα στην Πάρμα, στην Ιταλία, ένα μικρό οργανισμό που να συγκεντρώνει στοιχεία που προέρχονται από όλες τις χώρες της Ευρώπης και ουσιαστικά εστιάζει στην αξιολόγηση του κινδύνου. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα για το πώς συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Ένα παράδειγμα. Σήμερα το πρωί δημοσίευσε ο οργανισμός μας την ετήσια έκθεσή του για τα κατάλοιπα των παραστοκτώνων στα τρόφιμα. Το 97% των ε, τροφίμων που ελέγχθηκαν από τα κράτη-μέλη ήταν στα όρια είτε χωρίς καθόλου κατάλοιπα. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά τα τρόφιμα, η οποία τηρείται και είμαστε πολύ περήφανοι στην ΕΦΣΑ που παίζουμε αυτό τον πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν πρέπει όμως εδώ να μην είμαστε αυστηροί και να μειώσουμε την επαγρύπνησή μας σε κάθε περίπτωση μας ε, απασχολούν και τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές και θέλουμε να αξιολογήσουμε σωστά τους κινδύνους. Με την αλλαγή του κλίματος, με την αλλαγή στη συμπεριφορά των ε, καταναλωτών και με τις ραγδαίε τεχνολογικές αλλαγές στην ε, επιστήμη που αφορά την τροφική αλυσίδα και σε όλους αυτούς τους τομείς θα ήθελα να αναφέρω κάποια κατ λοιπά των ε, παρασιτοκτόνων, κάποιες ε, άλλες ε, επιδημίες, βακτήρια, κρίσεις στις οποίες προσπαθήσαμε στην ΕΦΣΑ να βρούμε αντι... αποτελεσματικές απαντήσεις και να αντιδράσουμε εγκαίρως. Και θα ήθελα επίσης να σας πω, όσον αφορά την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Υπάρχει εδώ συμφωνία ότι πρόκειται για ένα θέμα που απειλεί ιδιαίτερα τη δημόσια υγεία, η αντίσταση στα αντιβιωτικά. Και η ΕΦΣΑ από κοινού με το ECDC, την αρμόδια υπηρεσία για την πρόληψη των νόσων, κάναμε ελέγχους σε ζωοτροφές και σε τρόφιμα. Και περίπου 25.000 άνθρωποι πεθαίνουν στην Ευρώπη κάθε χρόνο διότι έχουν ε, προσβληθεί από βακτήρια τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντιβιωτικά σήμερα. Η κατάσταση είναι καλύτερη στις ε, βόρειες χώρες, στις νότιες χώρες της Ευρώπης και στην Ανατολική Ευρώπη. Η αντίσταση στα αντιβιωτικά είναι πολύ μεγαλύτερη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές ε, οι περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε όλα τα επίπεδα. Από το αγρόκτημα, από τον αγρό μέχρι στα επιστημονικά κέντρα. Και πολύ πρόσφατα δημοσιεύσαμε και μία έκθεση για να συμβουλεύσουμε τους πολιτικούς μας έτσι ώστε να πάρουν κάποιες αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο της μακροβιακής αντοχής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε τρόπο με διαφορετικές ε, ουσίες έτσι ώστε να μειωθεί αυτή η αντοχή. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει καλύτερη κατάρτιση, καλύτερη συνειδητοποίηση σε όλους τους εμπλεκόμενους και στους γεωργούς για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Άλλες ε, ασθένειες που πλήττουν ε, τα ζώα που ξεκίνησαν από την Αφρική, που σήμερα είναι παρούσες στη Μέση Ανατολή. Διάφορες δερματοπάθειες που έχουν φτάσει μέχρι και την Νότια Ευρώπη, την Ελλάδα, την Ανατολική Ευρώπη. Όπως παραδείγματο χάρη η οζόδης δερματίτης. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και σύμφωνα με τις ε, συμβουλές της ΕΦΣΑ είναι μια μαζική, ένας μαζικός ε, εμβολιασμός, κάτι που πιστεύουμε ότι θα είναι ο καλύτερος ε, τρόπος αντιμετώπισης αυτής της ασθένειας. Πιστεύω όμως ότι μόνο με τον τρόπο που δουλεύουμε και συλλέγοντα στοιχεία και δεδομένα από τα κράτη-μέλη θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα μπορούσα να σας δώσω και πολύ περισσότερα παραδείγματα. Αλλά θα σταματήσω εδώ. Ήθελα επίσης να μιλήσω και για τη σχέση μεταξύ της επιστήμης, των επιστημονικών δεδομένων και της λήψης αποφάσεων και της πολιτικής. Η επιστήμη αρχίζει και αντιμετωπίζει το θέμα των αξιών όταν τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα. Εμείς θέλουμε καταρχήν να γίνει μια κατανοητή επεξεργασία των επιστημονικών δεδομένων έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την λήψη αποφάσεων είτε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω εσεί πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και άλλα δεδομένα, όχι μόνο τα επιστημονικά. Υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα, πολλές φορές οι αξίες, η ηθική, η θρησκεία και όλα αυτά έτσι πρέπει να γίνονται από τη στιγμή βεβαίως που υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των επιστημονικών δεδομένων και της λήψης απόφασης. Καμιά φορά όμως υπάρχουν και εντάσεις μεταξύ των δεδομένων των επιστημονικών που παρέχουμε και αυτών των προσδοκιών ε, για τους πολιτικούς. Άλλα προσδοκούν οι πολιτικοί και άλλα συμπεράσματα βγαίνουν από τα επιστημονικά δεδομένα. Καμιά φορά λοιπόν εμείς γινόμαστε και η αποδιοπομπή, η αποδιοπομπή Και η γλυφωσάτη είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Ο οργανισμός μας α, εκπώνησε περίπου 40 συμπεράσματα για δραστικές ουσίες των λοιπασμάτων τα τελευταία χρόνια. 40! Και πέρασαν απαρατήρητα όλα αυτά τα συμπεράσματα και όλες οι σχετικές μελέτες κατά κανόνα. Πρόκειται για ένα στιβαρό κανονιστικό σύστημα που δεν στηρίζεται μόνο στο προσωπικό του οργανισμού μας, αλλά και σε 600 εμπειρογνώμονες από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Και είναι λίγο ηρωνικό αν εκπονήσουμε μία επιστημονική ε, μελέτη για τα την ταλοαμίνη, Μερικέ φορέ η επιστημονική κοινωνία, κοινότητα εγκομιάζει τον οργανισμό μα για το εξαιρετικό του έργο. Αλλά αν το ίδιο σύστημα, με του ίδιου ανθρώπου, με το ίδιο προσωπικό, με την ίδια διαδικασία, ε, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα για την γλυφοσάτη, για παράδειγμα, οι ίδιοι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών λέει στον οργανισμό μα, λάθο κάνετε, είστε μεροληπτικοί, είστε διεφθαρμένοι» και μάλιστα ένα ευρωβουλευτή δήλωσε δημόσια ότι, κατηγόρησε δημόσια την ΕΦΣΑ ότι σκοτώνει τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι πολύ επιλεκτική αυτή η αντιμετώπιση της ΕΦΣΑ, του οργανισμού μας. Και πολιτικά μπορεί να το κατανοήσω, αλλά διαρωτώ με πώς οι απλοί πολίτες θα εμπιστεύονται οργανώσεις όταν απαξιώνεται η φήμη τους και αμαυρώνεται η υπόλοιψή τους επειδή ακριβώς δεν συνάδει η μελέτη της με το πολιτικό πρόγραμμα του Α ή του Β πολιτικού. Πώ θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα, αν χαρακτηρίζονται από τα ίδια τα θεσμικά όργανα κάποια οργανισμοί κοινοτικοί ω αμεροληπτικοί, διεφθαρμένοι ακόμη χειρότερα. Θα πρέπει να, τηρήσουμε, να κρατήσουμε την προοπτική. Περίπου 500 ε, μελέτε επιστημονικέ το χρόνο εκπονούμε και μόνο λίγε φτάνουν στο φω τη δημοσιότητα και προσελκύουν την προσοχή του κοινού. Και γι' αυτό δημιουργούν μια δυσανάλογη φήμη για την ΕΦΣΑ. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Και αυτή είναι η έκκληση που σας κάνω. Σας θέλω παρακαλώ, σας εκλυπαρώ να έχουμε έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο ε, όταν μιλούμε για την επιστήμη και όταν μιλούμε και για πολιτική και για τις αξίες. Εγώ προσωπικά σας διαβεβαιώ ότι θα αξιοποιώ κάθε ευκαιρία για να έρχομαι στην Επιτροπή για να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και θα ήθελα ανακεφαλαιώνοντας να πω, ελπίζω να διευκρίνησα πόσο σημαντικός και σημαντικός είναι πόσο σπουδαίο και σημαντικό είναι ο ρόλο τη ΕΦΣΑ και για την αγροτική κοινότητα. Σα παρουσίασα κάποιε από τι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και θα να ακούσω και τι δικέ σα προσδοκίε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων και πώ μπορείτε και εσεί να συμβάλλετε στη διαμόρφωση του έργου μα. Γιατί όπω είπε και ο Πρόεδρο, θέλουμε να είμαστε περισσότερο στη διάθεσή σα ε, ε, για να στηρίξουμε το έργο σα, παρέχοντας σας ε, επιστημονικές γνωματεύσεις και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω και σε απορίες σας. Σας ευχαριστώ. Πολύ εμπεριστατωμένη και πολύ δυναμική η παρουσίαση που μας κάνατε. Θα περάσουμε τώρα στους ευρωβουλευτές, στα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Χόιμπουχ είναι η πρώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, ομιλία σας ε, μιλήσατε πάρα πολύ για το θέμα της εμπιστοσύνης, για την αξιόπιστη αξιολόγηση, για την εμπιστοσύνη εναντί των θεσμών. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να αξιολογήσουμε αυτούς τους θεσμούς και να υπάρχει εμπιστοσύνη, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι μελέτες ε, επιστημόνων, οι οποίες καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με τη βιομηχανία. Γιατί αν υπάρχουν μελέτες όπως έγινε προλίγου γνωστό η Μονσάντο, η μελέτη για τη γλυφοσάτα ανατέθηκε χωρίς όμως να αναφέρεται και να γνωστοποιείται το όνομα του ερευνητή. Αυτό λοιπόν ε, δεν είναι ένα μέτρο που να δημιουργεί εμπιστοσύνη και γι' αυτό ε, θα πρέπει κανείς να κατατάσει και τις ε, μελέτες. Αν θέλει κανείς ε, να δουλεύει τεκμηριωμένα, τότε δεν είναι δυνατόν να έχουμε μελέτες που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που είναι αυτονόητο είναι ότι αν θέλουμε πραγματικά να εμπνέουμε εμπιστοσύνη, τότε θα πρέπει ε, η προσφορά που υπάρχει να διακατέχεται από διαφάνεια. να μπορεί κανείς να ελέγχει τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της επιστήμης. Εσείς αναφέρετε μελέτες, οι οποίες βασίσεστε, αλλά κανένας ουδέτερος επιστήμονας δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα αυτά γιατί δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Και νομίζω ότι η ίδια η ΕΦΣΑ θα πρέπει να εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δουλεύοντας ε, με διαφάνεια και αποδίδοντας αξία στο ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διασύνδεση με τη βιομηχανία. Αυτό είναι από τα παλιά έτσι. Ξέρετε και εγώ έχω δύο γιους και οι δύο είναι επιστήμονες και δουλεύουν σε εταιρείε στη βιομηχανία Γερμανία ε, σπούδασαν πάρα πολλά χρόνια και ξέρουν πολύ καλά ότι όταν ε, ένας ε, κλάδος, μια εταιρεία πληρώνει και αναθέτει μια μελέτη, προφανώς το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη μελέτη είναι αρεστό στην εταιρεία. Κατά τα άλλα, πριν από 8 χρόνια δεν είχαμε το πρόβλημα με το τεοσύντε, είναι ένα είδος παρασίτου το οποίο ε, δεν υπήρχε τότε. Τώρα όμως υπάρχει το ΤΕΟΣΥΝΤ, κυρίως ε, στην Ισπανία. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι τι ακριβώς θα, κάνετε, ότι δεν είναι δυνατόν ε, να δεχτούμε ότι υπάρχει διασταύρωση με άγρια πανίδα. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά το πολύ παρακαλώ κάθε ομιλητής. Το πολύ. Λυπάμαι, αλλά θα σα διακόπτω. Σα ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη. Ο κύριο Άγγινου. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι δεν συνηθίζω να εκφράζω συμπάθεια για ευρωπαϊκού οργανισμού, αλλά για την ΕΦΣΑ θα το κάνω, γιατί επιστήμονε είστε, επιστημονικά πορίσματα εκδίδετε και άλλοι σα λένε «Α, σκουπίδια είναι αυτά που κάνετε, κάτι στραβό θα πρέπει να πηγαίνει με το υλικό αυτό, γιατί δεν, δεν δεν συμβαδίζει με το συμπέρασμα που περιμέναμε. Τι γίνεται, πού σταματήσαμε, καλά πήγαμε τη γλυφοσάτη, δεν βρήκατε τίποτα αρνητικό. Τη χρησιμοποιούμε εδώ και 40 χρόνια τη γλυφοσάτη και μάλιστα εγώ χρησιμοποίησα και συμπυκνωμένο πρωινό, προϊόν με γλυφοσάτη εδώ και πολλά χρόνια και ακόμη εδώ είμαι και υγιέστατος. Τι θα συμβεί λοιπόν στο μέλλον με τη γλυφοσάτη και τι, ποια θα είναι η χημική ουσία που το λόμπι τον οικολόγο θα καταδικάσει, ποια είναι στη, στον κατάλογό τους οι επόμενη. Επίσης, ε, ακριβώς επειδή είναι πολύ κακή η φήμη των φυτοφαρμάκων, αποθαρρύνεται ο κόσμος και δεν καταναλώνει φρούτα και λαχανικά. Αντί να καταναλώνει όμως χάμπουργκερ και πίτσες, καλύτερα φρούτα και λαχανικά να τρώει ο κόσμος. Αλλά με όλη αυτή τη διαφήμιση που γίνεται την αρνητική, ο κόσμος αποκαρδιώνεται. Επίσης με τα νεονικοτινοειδή. Πριν από λίγα χρόνια, δύο-τρία χρόνια ακούσαμε ότι είναι νευροτοξικά αυτά τα φυτοφάρμακα, βλάπτουν τις μέλισσες και σε μερικές περιπτώσεις ε, ε, στηριζόμαστε στην, ε, στη βαρότητα του φυτού για να καταπολεμήσει συγκεκριμένα παράσιτα. Δεν είναι δυνατό να μας λένε ότι οι ε, μέλισσες βλάπτονται και τώρα μας λέτε ότι δεν μπορούμε ούτε στα ζαχαρότευτλα να χρησιμοποιούμε τέτοια φυτοφάρμακα που περιμένουμε να ανθοφορήσουν μέχρι να τα, να τα μαζέψουμε. Επίσης, εκεί που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα είναι αυτό με τη, μικρο, είναι με τη μικροβιακή αντοχή. Και ελπίζω ε, η πράσινη, η, το πράσινο λόμπι να εμποδίσει τις προσπάθειές σας εκεί. Ο κύριος Δόρπον. Ευχαριστώ πολύ για τη θέση που πήρατε. Ήταν πάρα πολύ σαφής. Και βεβαίως ε, οι ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω είναι ότι αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι όσον αφορά τις παρασιτοκτόνα ιδιαίτερα για τα φυτά αυτά, για τα λαχανικά αυτά μεγάλων ε, εταιριών, μεγάλων επιχειρήσεων και τα επιστημονικά Ινστιτούτα δεν έχουν καμία σχέση με τις επιλογές αυτές. Ξέρουμε ποια είναι τα ανώτατα όρια για τα κατάλοιπα και από ό,τι ξέρω είναι ότι δεν είναι υπεύθυνη η ΕΦΣΑ, δεν επηρεάζει η ΕΦΣΑ άμεσα αυτά τα ανώτατα όρια, αλλά καλό θα ήταν να μας πείτε ότι η ΕΦΣΑ κάνει αυτό που έχει να κάνει. Δεν έχει νόημα εδώ αν απλώς για λόγους ε, επιστημονικούς, ο καθένας ε, πρεσβεύει τη δική του ιδεολογία και έχει τους δικούς του κανόνες. Ähm, ähm, Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ε, εδώ υπάρχει μια επικρατούσα άποψη ότι η ΕΦΣΑ οργανισμός αυτός ε, κάνει πολύ καλή δουλειά και μπορούμε να τον εμπιστευόμαστε. Ε, υπάρχουν βέβαια ε, κάποιες εναλλακτικές απόψεις. Αυτές, ξέρετε, ομαδούλες είναι που προσπαθούν για μικροπολιτικούς λόγους να προκαλούν και φόβο. Και νομίζω αυτά δεν πρέπει να τα υπερτιμούμε. Εγώ έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις αναφερθήκατε στην ε, οζόντι δερματίτιδα, σε αυτή την ε, ασθένεια και σε κάποιες άλλες βέβαια. Και θέλω να ρωτήσω, έχετε κάποιες πληροφορίες από αυτού. Νομίζω ότι οι εμβολιασμοί πήγαν πάρα πολύ καλά και αυτό είναι σημαντικό γιατί αν εξαπλώνεται αυτή η ασθένεια θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά στην Ευρώπη. Θέλω να ξέρω αν έχετε πληροφορίες από αυτού. Επίσης, ε, φτάνουν στα πια μας πολύ ανησυχητικές εκθέσεις σχετικά με το ούγκε 699, αυτή την ασθένεια ε, ότι έρχεται από την Αφρική προς την Ευρώπη. Έχετε κάποιες μελέτες επ' αυτού. Ε, έχετε κάποιες πληροφορίες ε, και σχετικά με το πρόβλημα με τους μήκητες οι μήκητες αυτοί έχουν πλήξει την Αφρική, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθούν στην Ευρώπη και θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον υπάρχουν ε, προτάσεις επ' αυτών. Ευχαριστώ. Κυρία Γιούσο. Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Τροφίμων που κάνει την παρθετική του εμφάνιση στην Επιτροπή Γεωργία. Γνωρίζω ότι ο ΕΦΣΑ έχει στιγματιστεί για πολλά θέματα, για έλλειψη ανε, ανεξαρτησίας, γιατί δεν είναι αρεστές όλα οι εκθέσει τα πορίσματα του ΕΦΣΑ. Εγώ όμως που είμαι αρμόδια για τη σχέση με τον ΕΦΣΑ, θεωρώ ότι είναι πραγματικά ανεξάρτητος οργανισμός και γνωρίζω τις επιστημονικές γνωματεύσεις που έχει κάνει και θεωρώ ότι είναι υψηλού επίπεδου όλες αυτές οι μελέτες και ξέρω ότι αναθεωρείτε την ε, πολιτική σας περί ανεξαρτησίας και κάνετε προσπάθειες να αυξήσετε τη διαφάνεια Ίσως αυτό έλειπε μέχρι στιγμής, όχι η αμεροληψία, αλλά η διαφάνεια. Και χαιρόμαστε για την προσπάθεια που γίνεται με τα υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας. Θα θέλαμε λοιπόν λίγες με περισσότερες διευκρινήσεις σε τι αναθεώρηση της πολιτικής σας γίνεται, ώστε να αποκαταστήσετε διαφάνεια ε, για να προβληθεί καλύτερα η ανεξαρτησία στην πολιτική σας. Ο κύριος Βαν Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διευθυντή της ΕΦΣΑ που είναι σήμερα εδώ και να κάνω και μία ερώτηση που αφορά τις απάτες και το κρέας αλόγων κυρίως στην Ισπανία. Διάφορα άλογα τα οποία πλέον δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον υπόδρομο βρέθηκαν τελικά στα κρεοπολία. Πρόκειται για μια απάτη και αναρωτιέμαι για άλλη μια φορά αν ο έλεγχος ε, στην τροφική αλυσίδα είναι αποτελεσματικός και θα θέλαμε να βρεθούν τρόποι έτσι ώστε να μην συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Έχετε κάποιες ιδέες τον Οκτώβριο του 2016 υπήρξε και ένας κανονισμός και εφαρμοστικές διατάξεις από μέρους της Επιτροπής, ιδιαίτερα για εισαγωγές ε, κρέατος από τρίτες χώρες και ίσως να υπήρχαν και κάποια ζώα που να μην είχαν καν εμβολιαστεί. Μπορείτε να, ασχολη... να μας πείτε πώς σκέφτεστε να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Η ταυτότητα των ε, ζώων τα άλογα παραδείγματος χάρη που βρίσκονται είτε ευρωπαϊκά είτε από τρίτες χώρες που τελικά βρίσκονται στην ε, παρασκευή τροφίμων. Μήπως όμως υπάρχει και στρέβλωση ανταγωνισμού και διαφορετική αντιμετώπιση για τα άλογα εντός και εκτός Ευρώπης. Πολύ ωραία, ε, πολύ σωστά τα είπατε. τον ε, έψα, το πιάξαμε ως οργανισμό για την αξιολόγηση κινδύνου. Δηλαδή, συνειδητά ε, θελήσαμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας σε επιστημονικές γνώσεις να πω το εξή. Θα έχω δύο ερωτήσει πολύ συγκεκριμένε. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξή. Νομίζω πολύ σωστά κάναμε να αποφασίσουμε να κρατήσουμε μικρό τον οργανισμό ΕΨΑ. Γιατί οι απαιτήσει ε, έναντι του οργανισμού αυτού είναι τόσε πολλέ που δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό ο υδροκεφαλισμό. Όσο μικρότερο οργανισμό, τόσο πιο αποτελεσματικά δουλεύει. Μερικές φορές ε, ε, κατηγορούν κάποιοι την ΕΦΣΑ ότι οι επιστήμονες δεν έχουν χρόνο ε, είναι πολύ απασχολημένοι. Μήπως μπορείτε εσείς να μας εξηγήσετε ποιος παίρνει πιο φάκελο από τους επιστήμονες για να διασφαλίζεται και η ανεξαρτησία τους. Η άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω έχει ήδη τεθεί αφορά στην στρατηγική αντιμετώπιση των επιδημιών που πλήττουν τα ζώα. Ε, είναι μια ερώτηση που γίνεται συνέχεια, γιατί στην Ευρώπη κάθε τόσα χρόνια αντιμετωπίζουμε τη γρήπη των πτηνών. Ε, αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα ε, σε μας στην Επιτροπή Γεωργίας και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κάποια συγκεκριμένη εντολή να διεξάγετε έρευνες που να αφορούν σε αυτές τις επιδημίες ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη από το 2013 περιορίσαμε κάποια μόρια από τα νεονικοτοειδή. Νεονικοτινοειδή. Καθότι υπήρχαν επιβλαβείς ε, επιπτώσεις ε, κυρίως στο περιβάλλον. Η ΕΦΣΑ, από ό,τι ξέρω, επανεξετάζει την επικινδυνότητα αυτών των ε, νεονικοτινοειδών. Και ενώ είχαν σταματήσει αυτές οι μελέτες, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για τα υπόλοιπα νεονικοτινοειδή που συνεχίζουν να υπάρχουν στην αγορά, καθώς και για την ε, βιομηχανική τους χρήση. Εγώ θα προτιμούσα να είχαμε θέσει το ερώτημα για την εντατική χρήση αυτών των ε, ουσιών και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε από αυτά το περιβάλλον. Ο κύριος Ανδρία, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εσάς κύριε Γενική Διευθυντά για την παρουσία σας και για τις παρατηρήσεις σας. Όπως ξέρετε είναι πολύ σημαντικός ο, ο ρόλος ο δικός σας στην διαμόρφωση των πολιτικών μας αποφάσεων και μέσω των δημόσιων διαβουλεύσεων είπατε ότι θα αναθεωρήσετε την πολιτική ανεξαρτησία σας. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος, ε, γιατί ε, είναι σημαντικό το διακύβημα της αξιοπιστίας ε, των επιστημονικών πορισμάτων του ΕΦΣΑ. Θα πρέπει και η και των πορισμάτων και η ανεξαρτησία και η αμεροληψία σας να είναι διασφαλισμένα. Επίσης, ίσως θα πρέπει να μπείτε και στη θέση του πολιτικού. Όταν έχουμε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που εκδίδουν αντιφατικές γνωμοδοτήσει, δεν είναι καθόλου εύκολη, εύκολη θέση μας, γιατί πρέπει να διαλέξουμε. Μπείτε λοιπόν και εσείς λίγο στη θέση μας. Και σίγουρα η ΕΦΣΑ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πολλό δε μάλλον τι τελευταίε εβδομάδε, μετά τι αποκαλύψει που έγιναν, ε, είχαμε κάποιες εξελίξεις, γιατί εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με τον αντίκτυπο της γλυφοσάτης στην ανθρώπινη υγεία και πολύ σωστά μιλήσατε για αξιοπιστία και σας ενδιαφέρει η αξιοπιστία του οργανισμού σας, αλλά ούτε και ο δικός μας ρόλος είναι εύκολος, γιατί έχουμε καθημερινά επαφές με τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, τι γίνεται με την επιστημονική αξιολόγηση που δεν θα ήθελα που δεν είναι να αφισβητήσω εδώ, και ως προς την ανάγκη των μελετών που συστανατέθουν περισσότερο οι δημόσιοι φορείς και όχι τόσο η βιομηχανία, γιατί όταν ο κλάδος σας αναθέτει την εκπόνηση κάποιων επιστημονικών μελετών, βλέπετε, βλέπετε ότι δεν είναι ορατά τα όρια μεταξύ του ε, δικαστή και του θύματος κατά κάποιο τρόπο, γιατί εκεί υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ενδεχομένω. Ο κύριος Χαϊτεμα. Ευχαριστώ κύριε Ούρλ για την παρουσίασή σας. Ε, συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε και τα υποστηρίζω. Σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή εντοχή, είναι πραγματικά μια τεράστια πρόκληση και ε, ευρωπαϊκός και παγκοσμίως και είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και με επιστημονικό τρόπο και θα πρέπει να σκεφτούμε νέε ιδέε. Επίση, κάνατε διάκριση μεταξύ επιστήμης και πολιτική. Θα πρέπει να παραμείνει σαφή αυτό ο διαχωρισμό μεταξύ τη επιστήμης και τη πολιτική. Για τα φυτοπροστατευτικά υλικά, για παράδειγμα, έχουμε ένα σύστημα που θα πρέπει να το καλλιεργούμε και να μας ικανοποιεί, γιατί είμαστε ευχαριστημένοι από το σύστημα που έχουμε μέχρι στιγμής. Και σε ό,τι αφορά τα νέο νοικοτινοειδή και τις, την περίπτωση αυτή για την ευρωτοξικότητά τους, όπως ξέρω, ο ΕΦΣΑ έχει κάποιες κατευθυντήρες γραμμές ε, που λαμβάνει υπόψη το θέμα των μελισσών. Στο Συμβούλιο βέβαια εκφράστηκαν αμφιβολίες για την ορθότητα αυτού του συστήματος. Πώς λειτουργεί αυτή η μελισσοκαθοδήγηση που έχετε συμπεριλάβει και τι γίνεται με το θέμα αυτό ως προς τη χρήση των νέων οικοτινόειδων. Η κυρία Γκυλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκτελεστικό διευθυντή του ΕΦΣΑ για την παρουσία του Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη και σκόπιμη παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας, γιατί πολλές συζητήσεις γίνονται και μερικές φορές αμφισβητείται και ο ίδιος ο ρόλος ε, του οργανισμού σας και η ορθότητα των επιστημονικών σας πορεσμάτων. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι Μερικές φορές ε, όταν ε, μιλούμε για αξίες ε, και για ηθική και διοντολογία, μερικές φορές αφιζητείται η επιστημονική ανάλυση. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τις αξίες και την ηθική τη διοντολογία με τα επιστημονικά συμπεράσματα. Γιατί αυτό συμβαίνει, ίσως όχι στην Επιτροπή μας, αλλά σίγουρα συμβαίνει πολλές φορές. Είναι έγκριτοι οι επιστήμονες του ΕΦΣΑ και το έργο τους πολύ αξιόλογο. Βέβαια, σκόπιμο θα ήταν να εμβαθύνουμε στα θέματα της διαφάνειας που επισήμανε κάποιος προλαλή σας. Και σίγουρα η μεγαλύτερη διαφάνεια θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το έργο του ΕΦΣΑ. Επίσης, δεν ξέρω αν σας αφορά, αλλά θα ήθελα να το σχολιάσω. Βλέπουμε ότι στις εισαγωγές από τρίτες χώρες η έλεγχη δεν είναι και πολύ αυστηρή. Είναι σχετικά επιπόλαιη. Για παράδειγμα, πώς μας διέφυγε ε, η εισαγωγή τέτοιων ποσοτήτων ε, νοθευμένου, αλλοιωμένου κρέατος από τη Βραζιλία και πώς είναι δυνατόν να εντόπισαν το σκάνδαλο οι βραζιλιάνικες αρχές και σε κανένα ευρωπαϊκό σύνορο, καμία τελωνιακή αρχή να μην εντόπισε αυτές τις παρτίδες με το σάπιο κρέας. Το ίδιο ε, συμβαίνει και με τα εσπεριδοειδή από την Νότια Αφρική. Και εκεί παρά ήταν ε, χαλαρή η έλεγχη στις εισαγωγές. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι να πείτε για το κατά πόσο είναι επαρκής ε, η έλεγχη στις εισαγωγές ή κατά πόσο επιδέχονται βελτιώσεις. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Σας ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομες. Καταρχήν, με ποιους μηχανισμούς θα εγγυηθείτε την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας των Τροφίμων και δεύτερον, με ποιους μηχανισμούς θα εγγυηθείτε την ανεξαρτησία κάποιων επαγγελματιών από τον κλάδο που φτάνουν ως εμπειρογνώμονες και στο δικό σας οργανισμό και πώς θα επιληθεί αυτή η σύγκρουση συμφερόντων. Ευχαριστώ κυρία Μίλλερ. Ευχαριστούμε πολύ ε, για αυτά που μας ε, είπατε. Εγώ εμπιστεύομαι τον ΕΦΣΑ και εκτιμώ πάρα πολύ και την πολύ καλή δουλειά που μας παρουσιάζεται. Βέβαια, για μένα που είμαι πολιτικός είναι απαραίτητο να γνωρίζω ότι μπορούμε ανα πάσα και στιγμή να καταφύγουμε σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα. Ε, Τώρα, ε, κατά πόσον μία μελέτη που πληρώνει η Μονσάντο είναι καλύτερη ή χειρότερη από μία μελέτη που έχει αναθέσει ο κλάδος προστασίας της φύσης, δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να μπληφτώ σε αυτά. Εγώ εκτιμώ προφανώς ε, την, ε, τον κλάδο προστασίας ε, της φύσης, πολύ πιο σημαντική αυτή από μια εταιρεία γιατί είναι πολύ πιο ανεξάρτητη και χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό ο οργανισμός ΕΦΣΑ και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ως πολιτική να έχουμε το θάρρος να αξιολογούμε τα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε με σαφήνεια. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Κατά πόσον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πορίσματα που προκύπτουν σε διάφορα κράτη. Έχω κατά νου μία μελέτη σχετικά με τις μέλισσες και τα νεονικοτονοειδή, μία μελέτη που έγινε στη Βαυαρία. Είχαμε μια συγκεκριμένη μονάδα όπου έγινε αυτή η μελέτη και θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα πορίσματα θα τα συμπεριλάβετε στις αξιολογήσεις σας ή όχι. Βεβαίω και με ενδιαφέρει η διαφάνεια, αυτό είναι ο σωστός δρόμος και νομίζω ο ΕΦΣΑ δεν έχει τίποτα να κρύψει. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο της διαφάνειας. Και για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας. Ο κύριος Ροπέ. Ačiū gerbiamas pirmininkė, Κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Το θέμα των κινητικά τροποποιημένων οργανισμών και η ελευθερία που έχουν τα κράτη-μέλη να τα καλλιεργήσουν ή όχι. Κάποιοι επέλεξαν ναι, κάποιοι επέλεξαν να μην το κάνουν. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη. Θεωρείτε ότι πρέπει να επεκταθεί αυτή η καλλιέργεια, ναι ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Κάποιοι ε, έλεγχοι που έγιναν όσον αφορά τα κατάλοιπα γλυφοσάτης στον ανθρώπινο οργανισμό έδειξαν ότι έχουν ξεπεραστεί κατά 20 ή 30 φορές αυτά στο νερό, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με το επιτρεπτό όριο. Το ίδιο και για τα τρόφιμα. Τώρα, όσον αφορά τον ε, πυρετό των... Ε, την πανόλη των χείρων, ξέρουμε ότι παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε και να εξαλείψουμε την νόσο αυτή. Δεν ξέρω βεβαίως ε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά ξέρω ότι στη Λετωνία, τη Λιθουανία και την Εστονία υπάρχουν αγροκτήματα που δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν την ασθένεια και εγκαταλείπουν την εκτροφή χείρων. Όσον αφορά τα εμβόλια και την καταπολέμηση αυτή της νόσου, δεν ξέρω, κανείς πια δεν ε, χρησιμοποιεί αυτά, αυτόν τον εμβολιασμό. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση αυτή της ε, νόσου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελαέρ. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δευθυνέου. Δεν είναι εύκολο να πάρει κανείς το λόγο μετά από τόσες πολλές ερωτήσεις. Εγώ πολύ θα ήθελα όταν πρόκειψε η κρίση της γλυφοσάτης να είχαμε αυτή την συζήτηση μαζί σας. Μας λέτε ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πολλοί σας κατηγόρησαν ότι δηλητηριάζετε τον κόσμο. Εγώ σαν συνεισηγήτρια ε, άκουσα κατηγορίες ε, όπως παραδείγματος χάρη ότι θα, θα δολοφονήσουμε τα παιδιά μας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύ παθιασμένη κατάσταση και είναι δύσκολο να πάρει κανείς ψύχρεμες αποφάσεις ε, σε αυτήν την ατμόσφαιρα και σε αυτό το κλίμα. Ο έλεγχος, η εκτίμηση από μέρους της ΕΦΣΑ είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται με ψυχραιμία για να μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε αποφάσεις. Όσον αφορά τα νικο και όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες να πάρουμε τις αποφάσεις μας βάσει επιστημονικών δεδομένων και με ψυχραιμία. Ο κύριος Ντές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ κύριε Διευθυντά που ήρθατε σήμερα εδώ. Ε, το ελάχιστο είναι να έρχεστε μία φορά σε εμά για να μπορούμε να συζητήσουμε. Πήξατε το αποτέλεσμα 97% το ε, τρόφιμα όπου ε, δεν διαπιστώθηκαν κατάλοιπα. Όμως υπάρχει το 3% που υπάρχουν ε, κατάλοιπα. Αυτό το 3% αφορά συγκεκριμένα τρόφιμα ή συγκεκριμένες περιοχές. Ίσως εξ αυτού μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα. Κατόπιν έγινε λόγος για την μικροβιακή εντοχή. Γνωρίζετε κατά πόσον αυτή αποδίδεται στην κτηνιατρική ή αν θέλετε και στην ιατρική που αφορά στους ανθρώπους, το δηλαδή προέκυψε αυτή η μικροβιακή εντοχή. Μετά είπατε κάτι άλλο, ότι ε, φτάνουν πάρα πολλές αιτιάσεις και κατηγορήσεις βάρους σας. Ε, μερικοί λένε σκοτώστε την εύσα. Εγώ διάβασα κάπου ότι ε, υπάρχει και μόμπινγκ σε παιδιά αγροτών ακόμα και ένας ε, πρόεδρος εκεί ενός αγροτικού συλλόγου είπε ότι τα έχει χάσει με αυτό τον εκφοβισμό των παιδιών των γεωργών. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ε, αυτά τα αποτελέσματα που έχετε, γιατί δεν τα παρουσιάζετε με ένα τέτοιο τρόπο, τουλάχιστον στους δασκάλους, έτσι ώστε να μην εκφοβίζονται τα παιδιά σε τέτοιο βαθμό που αναγκάζονται πολλέ φορέ και οι γονεί να εγκαταλείψουν τη Γεωργία γιατί δεν άντεχαν αυτόν τον εκφοβισμό των παιδιών. η Υπουργό ε, Γεωργίας, από ό,τι λέγεται, συνέβαλε στο να ενταθεί αυτός ο εκφοβισμός. Κατά τα άλλα όμως ε, πρέπει να ησυχάσουμε, να είμαστε και λίγο πιο ε, αισιόδοξοι. Έχουμε τον γιατρό, τον, τον γεωργό, τον δάσκαλο και τον επιστήμονα, κάτω-κάτω οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και οι πολιτικοί. Αυτή είναι η κατάταξη των πολιτών για το ποιον εμπιστεύεται περισσότερο. Το ότι υπάρχει αυτή η κατάταξη, εμένα πρέπει να σα πω, κάπως με καθησύχασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να πω ότι έχω να πω πράγματα, αλλά έχω και να μάθω και πράγματα. Όσον αφορά το ρόλο που διαδραματίζει ο ΕΦΣΑ, προφανώς και θέλουμε να σας εμπιστευόμαστε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω όμως ότι εξεπλάγει από αυτά που είπε η κυρία Μούλερ, ότι δηλαδή πρέπει να εμπιστευόμαστε τη Μονσάντο όπως ακριβώς εμπιστευόμαστε, αν θέλετε, μια επιστημονική ομάδα, περιβαλλοντική ομάδα μάλλον, που διεξάγει μια έρευνα. Δεν είναι έτσι, γιατί η Μονσάντο έχει στόχο πάνω απ' όλα ε, να αποδώσει χρήματα στους μετόχους με οποιοδήποτε τμήμα, τίμημα. Προφανώς λοιπόν οι μελέτες της Μονσάντο θα καταστήσουν σαφές ε, ότι τίποτα δεν μπορεί να τους ε, σταματήσει. Επίση, πρέπει να σας πω ότι με εκπλήσει και το εξής. Ξέρω έναν πατατοπαραγωγό και πολλές φορές τίθεται το δίλημα να δεχτεί κανείς ε, τη δηλητηρίαση ή τη λιμοκτονία. Ως γονιός πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ με τη χρήση αυτών των φυτοφαρμάκων. Όμως ε, μιλάω και στους γεωργούς και ξέρετε μου λένε αν δεν χρησιμοποιήσω αυτά τα φυτοφάρμακα δεν θα μπορέσω και εγώ να τρέψω τα παιδιά μου. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει μια κίνηση από τους πράσινους ευρωβουλευτές ε, και από έναν Ιρλανδό ευρωβουλευτή για το θέμα της γλυφοσάτης στην πρότασή του, ίσως τώρα να χρησιμοποιώ λάθος ονόματα, ο υπαριθμών 7 λένε ότι θέλουν να μηνύσουν την Μονσάντο γιατί έχει σκόπιμα στρεβλώσει τα στοιχεία για την γλυφοσάτη. Ε, το θέμα είναι ότι αν ισχύει αυτό πραγματικά ε, με ανησυχεί πάρα πολύ και από το πρίσμα της εμπιστοσύνης ε, η κοινή γνώμη ακούει αυτά, ακούει και τα άλλα αλλά ακούει και καταστάσεις όπου ο ΕΦΣΑ διαφωνεί με άλλους οργανισμούς ε, και υπάρχει ένα ερώτημα σε αυτή την πρόταση των Πρασίνων και του Ιρλανδού Ευρωβουλευτού ε, που λένε ότι ε, ο ΕΦΣΟ έχει πει να αποσυρθούν κάποιες μελέτες γι' αυτό θα πρέπει να αμφισβητήσουμε λιγάκι την αξιοπιστία του. Υπάρχει όμως η αναθεώρηση σχετικά με την γλυφοσάτη. Η γλυφοσάτη έχει αποδειχτεί ότι είναι επικίνδυνη και είναι καρκινογενής, καρκινογόνα. Ε, γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων, γιατί ο ένας οργανισμός λέει ότι πραγματικά ανησυχεί με τη γλυφοσάτη και εσείς λέτε ότι δεν ανησυχείτε και τόσο πολύ, όχι ιδιαίτερα, όσον αφορά την επικινδυνότητα της γλυφοσάτης. Σας ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω όμως κοιτάτε και λίγο το χρονόμετρο γιατί είπαμε όχι πάνω από δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Ευθύντα. Είμαι από αυτούς που πολλές φορές έχω επικρίνει την υπηρεσία σας όχι όσον αφορά την ουσία των εργασιών σας. Είστε πάρα πολύ χρήσιμοι για να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων μας. Είστε λοιπόν ένας πολύ χρήσιμος οργανισμός. Πριν από λίγα χρόνια με κάποιους συναδέλφους ήμασταν πάρα πολύ ε, επικριτική. Θυμάστε την κυρία Μανάτη, αν θυμάστε το βιογραφικό της, είχε λίγο τροποποιηθεί στον ιστότοπο της υπηρεσίας σας, καθότι ανήκε στο Ινστιτούτο, το Διεθνές Ινστιτούτο για την ε, ζωή πολύ ωραίος τίτλος, ε, εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ε, άλλων οργανισμών, αλλά και επιχειρήσεων όπως ε, την Μοσάντο και άλλων μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που παράγουν παρασιτοκτόνα και φυτοφάρμακα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν λάβατε κάποια μέτρα έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτησή σας από αυτό το Ινστιτούτο που έχει έναν πολύ βαρύγδουπο τίτλο αλλά που επηρεάζεται πολύ σημαντικά από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Μετά λοιπόν από την περίπτωση της κυρίας Μανάτη, που δεν ξέρω αν ήταν μοναδική περίπτωση, πήρατε κάποια μέτρα ανεξαρτησίας σε σχέση με το Ινστιτούτο αυτό, γιατί θυμάμαι ότι πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια είχαμε συζητήσει αυτήν την ε, περίπτωση. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, Διευθυντή ε, για το ότι ήρθε εδώ, είναι διαθέσιμος ακόμα και για τη σύγκρουση ε, μερικές φορές ε, πράγματι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες και από πλευράς μου ε, για την αποτελεσματικότητα της ΕΦΣΑ, αλλά παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι σέβομαι ιδιαίτερα άτομα που έχουν ιδιαίτερα προσόντα θα αναφερθώ σε κάτι που ε, φύγει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει τελικά να δώσει την μια ξεκάθαρη απάντηση. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω την ερώτηση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Χημικές Ουσίες, 15 Μαρτίου, ε, είπε ότι η γλυφοσάτη δεν μπορεί να θεωρείται καρκινογόνος ουσία, η γλυφοσάτη. Εκτός από αυτόν τον οργανισμό και ο ΕΦΣΑ είπε ότι το 2015 μέσα από, την, από το Διεθνή Οργανισμό περί Καρκινογενών Ουσιών ο οργανισμός αυτός ε, θεωρήθηκε η Γλυφωσάτη, ότι είναι καρκινογόνα. Υπάρχουν λοιπόν αποφάσεις από δύο οργανισμούς ε, που αυτές οι αποφάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να χρησιμοποιείται η γλυφοσάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμα 15 χρόνια. Αυτό που λείπει είναι μόνο ε, διότι εξετάζεται μόνο ένα μόριο με συγκεκριμένη ένωση και παραλείπονται πάρα πολλέ άλλε, με τι οποίε όμω η γλυφοσάτη εμφανίζεται στην αγορά. Εδώ πρόκειται για συνέργεια χημικών ουσιών. Με βάση λοιπόν τις ε, αποφάσεις ε, των δύο οργανισμών, όλα αυτά θα δοθούν σε ένα γερμανικό οργανισμό, ο οποίος ε, αναφέρεται και αυτός σε μια ειδική ομάδα που θα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς ε, των ε, ζυζανιοκτώνων. Το θέμα λοιπόν της γλυφοσάτης, αυτό το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο, εξετάστηκε από διάφορους επιστήμονες. Εγώ εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι όλα αυτά βρίσκονται σε, ε, σε σαφή αντίφαση με τα επιστημονικά πορίσματα. Εσείς ως διευθυντής του ΕΦΣΑ μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα έγγραφα εκείνα που βασιστήκατε ως ΕΦΣΑ για να αποφασίσετε σχετικά με την τοξικότητα της γλυφωσάτης. Η κυρία Σλάια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Διευθυντά, δυστυχώς δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα έγγραφα μόλις έφτασα. Έχω όμως μία ερώτηση για τις κάτω χώρες. Γιατί εμείς ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την νανοτεχνολογία, ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο του ΕΝΤ. Χρησιμοποιούμε νέα τρόφιμα και νέες τεχνικές και μέχρι στιγμής είχα καταλάβει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Πρόσφατα όμως Μία νέα οδηγία πλαίσιο για το είδωρ ε, υπευλήθη και εκεί ε, ε, ως επ' ευκαιρία αρχίζουν και ενισχύονται οι κριτικές. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι, πώς θα διαχωρίσουμε την αλήθεια από τις ανακρίβειες. Πρέπει να ενημερωθούμε γιατί πρέπει και η Επιτροπή Περιβάλλοντος να λάβει μια θέση. Ευχαριστώ κύριο Σφεγάν. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε να απαντήσω στην κυρία Ντελαέ. Εγώ είμαι λαϊκιστής ίσως, αλλά δεν είμαι, αν θέλετε, υπεύθυνο για όλα όσα συμβαίνουν. Δυστυχώς, σήμερα, αυτό που ζούμε είναι το αποτέλεσμα αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε θέματα περιβάλλοντος. Εδώ το θέμα της λασιμότητας, παραδείγματος χάρη. Δεν υπάρχει έλεγχος στην αλυσίδα παραγωγής, δυστυχώς. Και στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αρκετός αριθμός ελεγκτών. Το πιο σημαντικό όμως είναι η ετικετοθεσία. Από τον ε, Ιανουάριο του 2017 πρέπει να γίνονται έλεγχοι και μόνο ένα στα επτά προϊόντα έχει σωστή ετικέτα που αφορά την προέλευση, ιδιαίτερα όσον αφορά την προέλευση Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Υπάρχει πρόβλημα. Η προέλευση Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είναι ένα είδος κάλυψης απατών, παραδείγματος χάλιν για το κρασί ισπανικής προέλευσης, για το ελαιόλαδο, για το κρέας, το μποσχαρίσιο, παραδείγματος χάρη Και πιστεύω ότι αν γίνει καλύτερος έλεγχος και καλύτερη σήμανση, θα είμαστε σε θέση σήμερα να μιλήσουμε για προστασία, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Ο κύριος Χόισλινγκ. <clears throat> Κύριε Ουλ, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μας είπατε περίπου τα ίδια. Είχατε μία παρεμφερή ομιλία και τι κάνατε, στυλιτεύσατε δύο κόσμους. Την πολιτική αφενός και τους ανεξάρτητους επιστήμονες αφετέρου, τους οποίους δεν πρέπει και να εμπιστευόμαστε απόλυτα. Νομίζω τώρα κάπως πρέπει λιγάκι να τα διορθώσετε αυτά που είπατε, γιατί αυτή η ανεξάρτητη επιστήμη, ε, η επιστήμη έχει κάνει πολλά λάθη, Ντετετέ, Ατρατσίν, Λιντάν, Αυτά υποτίθεται ότι δεν δημιουργούσα κανένα πρόβλημα και μετά στο τέλο όμω τι διαπιστώθηκε. Διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν και τόσο ανεξάρτητη αυτή η ανεξάρτητη. Ξέρετε, αυτή η υποτιθέμενη ανεξάρτητη επιστήμη δεν υπάρχει και η πολιτική έχει ένα βασικό καθήκον ότι θα πρέπει να αποφασίζει ε, τι μπορεί να χρησιμοποιείτε και τι όχι. Ε, γι' αυτό λοιπόν το να δημιουργείτε εσείς ε, αυτή τη σύγκρουση, την ανεξάρτητη επιστήμη που υποτίθεται εκπροσωπείτε εσεί και από την άλλη η πολιτική, αυτό δεν είναι σοβαρό αυτή η διάσταση που προκαλείται. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος με τη δουλειά σας αν ε, τελικά πράγματι οι μελέτες ε, ήταν εξάρτητες. Ε, δεν είναι έτσι όμως. Και εσείς εξαρτάστε από το ότι πρέπει να ελέγχετε τις μελέτες της βιομηχανίας, αν έχουν νόημα, αν ε, ακολουθούν ε, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα δεν έχετε καμία δυνατότητα να ε, έχετε παντελώς ανεξάρτητες μελέτες, ούτε τα χρήματα έχετε, ούτε την υποδομή. Γι' αυτό τώρα μην εμφανίζεστε σαν να είσαστε παντελώς ανεξάρτητοι, εσείς απλά ελέγχετε τους ανεξάρτητους. Άρα δεν είστε και τόσο ανεξάρτητοι κι εσείς. Αν πραγματικά ήσασταν σε θέση να ελέγξετε κάτι καθαρά επιστημονικά και ανεξάρτητα, νομίζω ότι θα είχατε και τελείω διαφορετικέ απόψει. Και θα σας ε, εμπιστευόταν και διαφορετικά κοινή γνώμη. Όσον αφορά τα νεονικοτινοειδή, ε, πράγματι άλλοι θα σας ε, επικρίνουν, όχι εμεί. Υπάρχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Είπατε ότι το 97% των τροφίμων δεν επιβαρύνονται. Εγώ όμω λέω ότι το 3% είναι πάρα πολύ. Εσεί μπορείτε να συνδέσετε την μείωση τη βιοπικιλότητας με τη χρήση των φυτοφόρων. Τα Θα λέγατε άραγε ότι υπάρχει πράγματι σχέση ανάμεσα αυτά τα δύο ή είστε πεπισμένος για το αντίθετο. Ευχαριστώ κύριε Σμποβέ. Κύριε Ήρλα, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που σας βλέπω εδώ, γιατί εδώ και χρόνια συνεργάζομαι με τον ΕΦΣΑ και ευχαριστώ τον κύριο Ταραμπέλα που υπενθύμησε την υπόθεση Μπανάτη, γιατί Χάρη στην υπόθεση αυτή ξεκίνησε η ΕΦΣΑ μία προσπάθεια μεγαλύτερης διασφάλισης ανεξαρτησίας της και ε, θωράκης απέναντι στη σύγκρουση συμφερόντων. κάτι που δείχνει ότι έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Καταρχήν ε, είναι πολλές οι διαστάσεις αυτών των προβλημάτων. Το πρώτη διάσταση είναι το επιστημονικό θέμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μεθοδολογία σήμερα. Γιατί κάθε φορά που αξιολογείται ένα προϊόν, τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως βάση για την αξιολόγηση προέρχονται από την διαφερόμενη επιχείρηση. Το είδαμε και με τη Monsanto, με την Bayer και με άλλες επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα βασικά έγγραφα. Μετά ε, εμπλέκεται η Επιστημονική Επιτροπή που βλέπει αν υπάρχει βιβλιογραφία που συνάδει που απάδει από τα βασικά έγγραφα και υπάρχει κάτι μεροληπτικό στο γεγονός ότι τα βασικά έγγραφα προέρχονται από την ίδια την εμπλεκόμενη επιχείρηση, την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτή την εξάρτηση, γιατί από τη στιγμή που τα βασικά έγγραφα είναι μεροληπτικά και προέρχονται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, πώ θα διασφαλίσουμε μετά την διόρθωσή του στη συνέχεια. Θα συνεχίσουν να είναι μεροληπτικά. Δεύτερο επίπεδο. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι θέλουμε να είναι πιο ανεξάρτητος οργανισμός. Και εσείς εγκύψετε και στο εσωτερικό του οργανισμού στο θέμα αυτό. Αλλά ο μόνος τρόπος για να είναι ανεξάρτητος οργανισμός είναι να είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος οικονομικά. Αν δηλαδή θέλουμε πραγματικά έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό, ανεξάρτητο από τον κλάδο, θα πρέπει στα πλαίσια του κοινοτικού προϋπολογισμού να πρικοδοτήσουμε τον οργανισμό με κονδύλια ε, τουλάχιστον διπλάσια από αυτά που έχει σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να πετούμε ανεξαρτησία χωρίς να προβλέπουμε τα κατάλληλα κονδύλια για να τη διασφαλίσουμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε ξυπνάδα, ευφυία και για να προσπίσουμε την ανεξαρτησία και να προστατεύσουμε τον ΕΦΣΑ θέλουμε επαρκή κονδύλια. Έτσι πραγματικά θα έχουμε εμπειρογνώμονες σε κάθε επιμέρους κλάδο που θα είναι πραγματικά ανεξάρτητοι, που δεν θα χρειάζεται να απασχολούνται και αλλού και έτσι θα διασκεδάσουμε οποιαδήποτε αφιβολία περί σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θέλουμε λοιπόν περισσότερα χρήματα για τον ΕΦΣΕ. Είναι η μόνη λύση για την ανεξαρτησία του οργανισμού. Δεν έχουμε άλλους αγορητές στον κατάλογο, οπότε θα παρακαλέσω τον Γενικό Διευθυντή να απαντήσει. Σας θερμοπαρακαλούμε να περιοριστείτε σε ένα τέταρτο αν γίνεται. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Σε 15 λεπτά να απαντήσω σε τόσες πολλές ερωτήσεις είναι μεγάλη πρόκληση. Θα ξεκινήσω όμως με τον κύριο Μποβέτα τελευταία λόγια του. Περισσότερα χρήματα για την ΕΦΣΑ. Μα όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας για τον οποίο είστε αρμόδιοι, θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο θέμα της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και τα δεδομένα. Πολλοί ανέφεραν το θέμα των δεδομένων. Ο κανονισμός αυτού του κοινοβουλίου είναι αυτός που υποχρεώνει κάποιον που θέλει να πάρει άδεια να υποβάλει δεδομένα τα οποία θα επιτρέψουν σε αυτόν ο οποίος ελέγχει τον κίνδυνο να αποφανθεί. Και αυτό ισχύει για τα πάντα, για τα φυτοφάρμακα, για τις ουσίες και για τα παραστοκτόνα. Και α, μπορεί κάποιος να επικρίνει αυτό το γεγονός, αλλά πρόκειται για κανονισμό, για νομοθεσία. Αν λοιπόν ε, κάτι πρέπει να αλλάξει, εδώ εσείς είστε οι αρμόδιοι. Χρειαζόμαστε τις νομοθετικές ε, αρχές, δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, που να αλλάξουν τους κανόνες υπό τους οποίους γίνονται οι διαδικασίες, οι έρευνες και ο έλεγχος στην Ευρώπη. Και βεβαίως εδώ έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Πρόκειται για μια μεθοδολογία η μεθοδολογία αυτή δεν έχει εφευρεθεί από τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για πρότυπα που έχουν οριστεί από τον ΩΣΑ. Ο ΩΣΑ είναι αυτός που καθορίζει τις κατευθύνες γραμμές για να γίνουν, παραδείγματος χάρη, πειράματα στα ποντίκια και πρόκειται για πειράματα είτε είναι σε εργαστήρια είτε είναι σε ε, ακαδημαϊκά ιδρύματα που γίνονται βάσει της ίδιας ε, μεθοδολογίας. Αν όμως μου πείτε ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον, στο αποτέλεσμα μιας έρευνας, επειδή την έχει παραγγείλει μια επιχείρηση, αυτό πλήττει την αξιοπιστία κάθε οργανισμού. Εμείς όμως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κανονισμό. Εμείς ε, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε όλα τα δεδομένα που μας υποβάλλει αυτός που ζητά την επιστημονική μελέτη, να στραφούμε προς όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που υπάρχουν στην ε, ε, διεθνή αν θέλετε, επιστημονική γραμματεία και κατόπιν να διεκπαιρεώσουμε την έρευνά μας. Σήμερα, παραδείγματο χάρη, στην ε, Αμερική γίνεται μία μελέτη για την τοξικότητα της βυσφενόλης. Και μία μελέτη Μία, αυτή η μία και μοναδική μελέτη στοιχίζει εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μιλάμε εδώ μόνο για 5 εκατομμύρια αύξηση του προϋπολογισμού μας, αναφερόμαστε σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια. Και αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό και πρόκειται για αυτούς οι οποίοι ζητούν μελέτες και οι οποίοι θα είναι σε ε, θέση να την χρηματοδοτήσουν, να την πληρώσουν. Εμείς πιστεύουμε, είμαστε πεπισμένοι θα έλεγα, ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε, να αξιολογήσουμε μελέτες όποιος και να τις έχει παραγγείλει και ζητήσει. Θα πρέπει λοιπόν και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο σύστημα αυτό, το οποίο σύστημα είναι το ίδιο όπου και αν γίνονται οι μελέτες. Εάν θέλετε να το αλλάξετε, εσείς μπορείτε να το αλλάξετε. Όσον αφορά τώρα την ανεξαρτησία των ε, εμπειρογνωμόνων μας, πόσο ανεξάρτητη είναι. Έχουμε, όπως σας είπα, 350 υπαλλήλους. Πρέπει όπως ξέρετε, να δηλώνουν τα συγκεκριμένα τους συμφέροντα και αυτό γίνεται σε ετήσια βάση. Έχουμε άτομα που εργάζονται με πενταετής συμβάσεις, δεν έχουμε υπαλλήλου και χρησιμοποιούμε και εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια πάρα πολύ έξυπνη κατά την άποψή μας απόφαση του νομοθέτη, διότι όταν εργαζόμαστε παραδείγματος χάρη για έντομα για μια συγκεκριμένη παραδείγματος χάρη κατηγορία τροφίμων, ζητάμε από τους εμπειρογνώμονες του ενδιαφερόμενου κράτου μέλους να μας παρέχουν στοιχεία. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία τους. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια, ανεξαρτη... μια πολιτική ανεξαρτησίας. Όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί μας πρέπει να κάνουν δηλώσεις συμφερόντων. Έχουμε 8.000 τέτοιες δηλώσεις το χρόνο για 35.000, αν ε, θέματα που εξετάζουμε κάθε χρόνο. Είναι μια πολύ σημαντική, αν εργασία για μας, αυξάνει το φόρτο εργασίας μας, αλλά το κάνουμε διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των ε, ε, μελετών μας και των συνεργατών μας. Αν κοιτάξετε το πρόγραμμα εργασιών μας, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε εταιρικέ σχέσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε και με τον ιδιωτικό τομέα και με τις επιχειρήσεις. Ε, και οι επιστήμονες το ίδιο. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει η έρευνα, δεν μπορεί κάποιος να έχει σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας. Διότι αν πεις ότι από τη στιγμή που χρηματοδοτείται μία μελέτη, μία έρευνα και από τις επιχειρήσεις και από τη βιομηχανία, καταλαβαίνετε ότι δεν θα προχωρήσουμε ούτε στην έρευνα ούτε στις μελέτες μας. Η Ευρώπη δεν θα είναι ανταγωνιστική. Η πλήρης ανεξαρτησία είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άλλο είναι η σύγκρουση συμφερόντων και άλλο είναι να διαλέξουμε εμπειρογνώμονες, επιστήμονες οι οποίοι έχουν εργαστεί στην πραγματική αγορά και γνωρίζουν τα πραγματικά προβλήματα. Και βεβαίως η πολιτική μας είναι αυτή που εσείς έχετε αποφασίσει, προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε, κάνουμε δημόσιες διαβουλεύσεις και μάλιστα μία βρίσκεται εν εξελίξη για τη νέα πολιτική μας τα θέματα ανεξαρτησίας. Χρειαζόμαστε και τη δική σας συνεισφορά και τη δική σας συμβολή έτσι ώστε να βελτιωθεί η νέα μας πολιτική ανεξαρτησίας. Θεωρούμε ότι είμαστε εξαιρετικά ανεξάρτητοι, χωρίς να μπορώ εδώ να πω ότι είμαστε, είναι τέλεια αυτή η πολιτική. Κάθε μέρα προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε από τη μία την αξιοπιστία των επιστημόνων μας, των εμπειρογνωμόνων μας και από την άλλη την ανεξαρτησία τους από τις επιχειρήσεις. Όλα όσον αφορά τη διαφάνεια βρίσκονται στην, στον ιστότοπό μας. Και αυτό ισχύει και για τη μελέτη για τη γλυφοσάτη. Πολλοί μας λένε γιατί δεν δημοσιεύετε όλες αυτές τις μελέτες που χρησιμοποιείτε για να γνωμοδοτήσετε. Καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε μία μελέτη θεωρεί ότι είναι δική του πνευματική διοκτησία. Και αυτό προστατεύεται στην Ευρώπη. Αυτό που δεν θέλουν οι επιχειρήσεις είναι ένας ανταγωνιστής τους να πάρει αυτή τη μελέτη και να πάει στην Κίνα ή στη Βραζιλία κάπου αλλού, να πάρει άδεια διάθεση στην αγορά με μια μελέτη η οποία χρηματοδοτήθηκε από άλλη επιχείρηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πρέπει να εξισορροπήσουμε την διαφάνεια αλλά και την υποχρέωσή μας να σεβαστούμε τα πνευματικά δικαιώματα. Τα πράγματα δεν είναι λοιπόν άσπρα ή μαύρα. Πρέπει κάθε φορά να πάρουμε μία απόφαση, να βασιστούμε στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηριού. Υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πολύ πρόσφατα μάλιστα υπήρξε και μία απόφαση για την σύμβαση του Άρχους που άλλαξε τα πράγματα. Πολύ πρόσφατα μάλιστα δημοσιεύσαμε και μία μελέτη με όλα τα δεδομένα για τη γλυφωσάτη μετά από αίτημα τεσσάρων ευρωβουλευτών. Αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε και να γίνουν γνωστά όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα. Και ξέρετε ότι αυτές οι μελέτες μπορούν να, από τη στιγμή που δημοσιεύονται, να αναπαραχθούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που μας επιτρέπει όπως ξέρετε, ο κανονισμός. Δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε ούτε στην ιστοσελίδα μας, ούτε πουθενά, δεδομένα τα οποία δεν μας ανήκουν. Έχω ακόμα λίγα λεπτά. Πολύ σύντομα, αφήστε με να κοιτάξω κάποιες από τις ερωτήσεις τις οποίες δεν απάντησα. Κύριε Ντόρφμαν, είπατε αν είναι χρήσιμο να πάμε σε κατώτερα όρια ακόμα όσον αφορά τα κατάλοιπα. Για μένα τα όρια τα οποία έχουμε θεσπίσει είναι όρια ασφάλειας ε, και οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτά τα όρια είναι τρόφιμα το οποίο είναι ασφαλή. Οτιδήποτε ξεπερνάει τα όρια βεβαίως σίγουρα δημιουργούνται ερωτηματικά. Για μας οτιδήποτε είναι κάτω από το όριο πάντως δεν έχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας. Κυρία Αγιούζο, μιλήσατε για την ανεξαρτησία. Προσπαθούμε και εμείς να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι προτάσεις και οι συμβουλές σας είναι καλοδεχούμενες. Επίσης, όπως σας είπα, υπάρχουν και δημόσιες διαβουλεύσεις, τις οποίες επίσης μπορείτε να συνεισφέρετε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, όσον αφορά τους επιστήμονες που χρησιμοποιούμε, συνεργάζονται με πανεπιστήμια, με ερευνητικά κέντρα, με Ινστιτούτα στα κράτη-μέλη και πληρώνονται από αυτά. Αυτό που πολλές φορές ακούμε όταν ψάχνουμε για πολύ καλούς επιστήμονες είναι ότι βεβαίως μπορούμε να έρθουμε να εργαστούμε για σας, αλλά χρειαζόμαστε πολύ ψηλότερους μισθούς, 1000 ευρώ την ημέρα δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτά τα ποσά. Βασιζόμαστε λοιπόν σε άτομα που εργάζονται, πληρώνονται από τα κράτη-μέλη και 50 ημέρες το χρόνο εργάζονται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε εθελοντική βάση. Καταλαβαίνετε όμως ότι με την κρίση τα κράτη-μέλη αρνούνται πλέον να μας διαθέσουν τους καλύτερους επιστήμονες τους. Το ευρωπαϊκό μοντέλο λοιπόν είναι ένα πολύ έξυπνο μοντέλο, το οποίο όμως έχει και τα αδύναμα στοιχεία του. Καταλαβαίνετε ότι τα κράτη-μέλη διαθέτουν τους καλύτερους επιστήμονές τους ως ένα βαθμό για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και αυτό για μένα είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για το άμεσο μέλλον. Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τους καλύτερους επιστήμονες χωρίς να τους πληρώνουμε, χωρίς να τους παρέχουμε πολύ σημαντικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Χρειαζόμαστε πολιτική στήριξη από μέρους των κρατών μελών και από μέρους του Κοινοβουλίου. Για τα νεονικοτινοειδή τώρα έγιναν κάποιες ερωτήσεις. Το 2013 υπήρξε η απαγόρευση και μας ζήτησε η Επιτροπή κάποια επιπλέον δεδομένα που να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που διαθέτουμε για τα νεονικοτινοειδή. Αυτό που σήμερα κάνουμε είναι μια επανεκτίμηση για, τα, για τις ουσίες αυτές που θα δημοσιευθεί το Νοέμβριο του 2017 με νέα συμπεράσματα για τα νεονικοτινοειδή και τη χρήση τους στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο για την ε, μέλησο καθοδήγηση, καθοδήγηση, Guidance, ε, που εξετάσαμε με τα κράτη-μέλη το 2013 και 2014, δεν έχει ε, γίνει πλήρω εκτός ακόμη από τη μόνιμη επιτροπή λόγω των επιφυλάξεων κάποιων κρατών μελών. Πάντω, χρησιμοποιούμε αυτέ τι νέε κατευθυντήριε γραμμέ κατέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στηρίζεται στα νέα εγγραφά κατευθυντήριο γραμμών. Έχω πολλά να προσθέσω, αλλά εξαντλήθηκε ο χρόνος που μου δώσατε. Καταρχήν, ε, είμαι στη διάθεσή σας να αποστείλω και γραπτός ε, απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν πρόλαβα να καλύψω. Θα λάβετε και γραπτή απάντηση. Πολύ ευχαρίστως όποτε θέλετε να έρχομαι στην Επιτροπή σας, αλλά και διμερώς μπορούμε να συζητούμε λεπτομέρειες και πολύ ευχαρίστω να έρχομαι μια φορά το χρόνο στην Επιτροπή σας για να έχουμε μια τακτική ανταλλαγή απόψεων. Και ως συνήθως περισσότερο μαθαίνουμε από τις ερωτήσεις σας παρά από τις απαντήσεις μου. Χαίρομαι λοιπόν για την πλειάδα των ερωτήσεων που επευλήθησαν και σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δώσατε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσία σας, κύριε Διευθυντά. Και ήταν πραγματικά τεράστιο το φάσμα των ερωτήσεων και των παρατηρήσεων. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν απαντήθηκε η απορία του και θα ήθελε να ρωτήσει κάτι επιπλέον, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Δεν βλέπω όμως ε, συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ο διευθυντής μας έδωσε την ευκαιρία. Α, συγγνώμη. Το περίμενα, φυσικά το περίμενα. Ε, αν, είναι δυνατόν ο κύριος Άγνιο θα χάσει ευκαιρία να θέσει ερώτηση. Οι κύριοι Χόισλιν και Φλάνεγκαν είχαν περίπου τρία λεπτά. Έχω και άλλη ερώτηση για τα νεονικοτινοειδή. Γιατί δεν κάνετε δοκιμές σε κλίμακα αγροκτημάτων, γιατί θα θέλαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μερικές περιοχές να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες όχι. Οπότε να εμπλέξουμε και τους μελισσοκόμους για να δούμε πού είναι μεγαλύτερη θνησιμότητα των μελισσών δεν έχει γίνει σε μεγάλη κλίμακα ακόμη. Καλό θα ήταν από αυτό να διδαχθούμε. Και προσπαθώ να πείσω, ε, προσπάθησα να πείσω τον ε, Υπουργό Γεωργία να το κάνει, γιατί πραγματικά δοκιμέ στα χωράφια θα μα πούν πολύ περισσότερα από ότι οι εργαστηριακέ δοκιμέ που γίνονται από επιστήμονε μόνο, σε κλειστέ πόρτε. Ο κύριο Γιάρ. Και εγώ να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση για τα νεονικοτινοειδή, γιατί τα έχω χάσει. Έχω μπερδευτεί. Υποτίθεται υπάρχει μια μελέτη, αλλά δεν τη δημοσιεύεται. Και παρόλα αυτά η Κομισιόν ε, φαίνεται ότι έχει λάβει κάποιε αποφάσει. Ε, θέλει να απαγορεύσει τα νεονικοτινοειδή νεονικοτονοειδή. Κάπως δεν ταιριάζει αυτό. Ε, θα πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή υπάρχουν πορίσματα που δεν δημοσιεύονται, όμως η Κομισιόν λαμβάνει αποφάσεις. Αυτό μοιάζει με πολιτική Κρεμλίνου, που το Κρεμλίνο αποφασίζει χωρίς να λέει τίποτα. Τώρα τι γίνεται, έγινε μελέτη, υπάρχουν πορίσματα. Γιατί η Κομισιόν δεν τα δημοσιοποιεί και πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν με μία μη δημοσιοποιημένη μελέτη ήδη να προχωράει σε αποφάσεις. Μάλιστα. πολύ ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις για τις μέλησες και θα έχουμε όλο και περισσότερες απορίες για αυτό το θέμα, οπότε θα ήθελα όταν μας στείλετε και γραπτός κάποιες πληροφορίες να έχετε περισσότερες, ε, περισσότερα στοιχεία για τις μέλησες, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Μάλιστα για τα νεονικοτινοειδή, όπως ε, θα φαντάζεστε δεν είμαι σε θέση εδώ να εκπροσωπήσω, να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο του 2016 δημοσιεύσαμε τρεις εκθέσεις για επιβεβαιωτικά στοιχεία και επιβεβαιώσαμε τον κίνδυνο που υπάρχει για τις μέλησες από τις ουσίες αυτές. Η πλήρης επαναξιολόγηση θα υποβληθεί το Σεπτέμβριο του 2017. Σε ό,τι αφορά τι μέλισσε, εδώ και πολλά χρόνια ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Τροφίμων ασχολήθηκε με την υγεία των μέλισσών και μα ενδιαφέρει μια σφαιρική προσέγγιση για του στρεσογόνου παράγοντε που επηρεάζουν την επιβίωση των κυψέλων. Ε, ε μπορεί να είναι η βακτήρια, παράσιτα, ε, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν επιμέρους παράγοντες, αλλά μια σφαιρική εξέταση των στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζει την επιβίωση των μελισσών. Και μάλιστα έχουμε ένα σημαντικό εργαστήριο στη Γαλλία με το οποίο συνεργαζόμαστε. Έχουμε ε, συνεργασία και με μελισσοκόμους και είμαστε στη διάθεσή σας για να δημιουργήσουμε μία ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για τις μέλισσες, αν συμφωνείτε κι εσείς, ώστε να υιοθετήσουμε πραγματικά μια πολυδιάστατη, πολυκλαδική και σφαιρική προσέγγιση, γιατί από μαθηματική και επιστημονική άποψη δύσκολο είναι να καταλήξουμε σε μοντέλα ε, για το πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά των μέλησών. Πάντως και εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα και πολύ ευχαριστώ να σας ενημερώσουμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επιβίωση των μέλησων και στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε και πάλι τον εκτελεστικό διευθυντή του ΕΦΣΑ για την παρουσία του. Και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 5 ε, που αφορά τις κλιματικές αλλαγές, εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Και όπως είπα θα ακούσουμε την παρουσίαση της μελέτης, ευχαριστώντας και πάλι τον κύριο Ούλ, ε, της ε, την προσή τη μελέτη που ζητήσαμε για τη συνέπειες των πολιτικών στο τομέα της αλλαγή του κλίματος ε, για τη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέχεια της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών COP21 του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ε, το τμήμα 2 της, ε, ε, ε, της πολιτικής εκπονήθηκε, ε, από το τμήμα μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Γεωργία αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια της πολιτικής ε, ε, μετριασμού των κλιματικών αλλαγών, της COP21 δηλαδή. Και θέλουμε να δούμε τις συνέπειες των συμφωνιών της COP21 για τη Γεωργία και ποιες θα είναι οι προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές ε, πολιτικές και πώς θα επηρεάσουν αυτές τη γεωργία. Πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί η μελέτη αφορά κυρίως το ρόλο της κοινή γεωργικής πολιτικής και το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η ΚΑΠ μετά το 2020 ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προσπάθεια μείωσης ε, των αερίων του θερμοκηπίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονές μας, την κυρία Κάλι Χάρτ και τον κύριο Μπεν Άλεν από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως ήθιστε θα ακούσουμε πρώτα τους καλεσμένους εμπειρογνώμονες και μετά τους ευρωβουλευτές. Έχετε 20 λεπτά στη διάθεσή σας. Πρώτα θα μιλήσει η κυρία Χάρτ. Δεν ξέρω αν θα εξαντλήσετε εσείς το 20 λεπτό ή θα το μοιραστείτε με τον κύριο Μπεν Άλεν. Και πώς θα απαντήσετε μετά σε ερωτήσεις. Αυτό εξαρτάται από εσά πώς έχετε συνεννοηθεί. Πάντως μαζί έχετε ένα 20 λεπτό. Καλώς ήρθατε και περιμένουμε την παρουσίαση της μελέτης σας. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, we will actually do this in a slightly... ΕΕΕΕ Αλλιώ θα τα κάνουμε, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω εγώ και μετά θα δώσω το λόγο στην Κέλλη για να κάνει το δεύτερο σκέλο. Σα ευχαριστούμε πολύ που μα δεχτήκατε σήμερα εδώ για να σα παρουσιάσουμε την έκθεσή μα. Ε, ελπίζω ότι θα έχετε κι εσεί ε, κάποιο αντίγραφο. Έχει πάρα πολλέ λεπτομέρειε, αυτή η μελέτη ε, με πολλές επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα από την συνεδρίαση COP21 και από τη Συμφωνία των Παρισιών, Όπω επίση και από τι πρόσφατες πρόσφατες προτάσεις Κομισιόν. Η μελέτη μας εξετάζει το ρόλο της ΚΑΠ στο να υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορεί να γίνει μετά το 2020. Όπως σας είπα λοιπόν, ε, θα εξετάσω εγώ ε, τα δύο πρώτα σκέλη της παρουσίασής μας, της μελέτης μας. Είναι η ε, σχέση ανάμεσα στη γεωργία και το κλίμα, επιπτώσεις στο, της γεωργίας στο κλίμα και τα Νάπαλιν. Επίσης θα εξετάσουμε και ε, το πώς ακριβώς η γεωργία παίζει ρόλο και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Και κατόπιν η συνάδελφός μου θα μιλήσει για το ρόλο, τον κλιματικό ρόλο της ΚΑΠ και για τις προοπτικές του μέλλοντος. Όσον αφορά λοιπόν την ανηλενδυσία ανάμεσα στην γεωργία και το κλίμα, η ίδια η γεωργία ως τομέας είναι τομέας παραγωγής. Βασίζεται και επηρεάζεται από το κλίμα με πάρα πολλού τρόπου. Ε, και αυτό ισχύει είτε αλλάζει το κλίμα είτε ή όχι. Ε, το μόνο που χρειάζεται είναι να δει κανεί πώς έχουν κατανομηθεί τα διάφορα συστήματα παραγωγής και διανομής ε, στην Ευρώπη. Έχουμε τι βόρειες χώρες με μικρότερες περιόδους ανάπτυξης, με πολλές βροχές και μετά μπορούμε να δούμε στο νότο έχουμε ξηρασία, Βλέπουμε λοιπόν ε, ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές ε, στο κλίμα. Οι ε, χειμώνες είναι λίγο πιο ήπιοι. Υπάρχουν όμως αλλαγές και στο καλοκαίρι. Εξάλλου βλέπουμε ότι αλλάζει και η διαθεσιμότητα των υδάτων. Ως εκ τούτου ε, διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις, βλέπουμε να υπάρχουν έντονες πλημμύρες ε, σε πάρα πολλές περιοχές και βλέπουμε να υπάρχουν περισσότερες θύελες, ε, κίνδυνος πυρκαγιάς, αυτό σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Όσον αφορά τώρα ε, τις ε, καλλιέργειες διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι επιβλαβείς οργανισμοί που μετακινούνται στην Ευρώπη. Όσο ε, πιο ζεστοί γίνονται οι χειμώνες δεν παγώνουν οι επιβλαβείς αυτοί οι οργανισμοί και αρχίζουν λοιπόν να επηρεάζουν τα συστήματα καλλιέργειας. Όλα αυτά είναι ένα είδος φυσικής αντίδρασης. Οι γεωργοί επηρεάζονται και οι γεωργοί επηρεαζόταν ανέκαθεν από το κλίμα, όμως το γεγονός ότι αλλάζει το κλίμα. Ε, σημαίνει ότι και οι γεωργοί καλούνται πλέον να ανταποκριθούν σε αυτές τις κλιματικές ε, εναλλαγές. Στη γεωργία, επιπτώσει στη γεωργία από το κλίμα, βλέπουμε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι που το αντιμετωπίζουμε. Ο πρώτος είναι ότι η γεωργία ε, προκαλεί ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέσα από τις αλλαγές ε, του τρόπου με τον οποίο καλλιεργείται η γη λόγω του μεθανίου και λόγω και των, της χρήσης της ενέργειας στη γεωργία. Αυτό που είναι μοναδικό όμως στη γεωργία σε ολόκληρη την οικονομία είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να περιοριστούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα με τη δέσμευση του άνθρακα, παραδείγματο χάνει στη βιομάζα. Δηλαδή υπάρχουν επιπτώσεις και στη δέσμευση του άνθρακα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ως απάντηση της Γεωργίας για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η Γεωργία διαδραματίζει ρόλο στο να περιστούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα και σε άλλους ε, τομείς, ε, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βιομάζα, επίσης να αλλάξουν και οι υποδομές, να υπάρχουν ανεμογεννήτριες, ε, παραδείγματο χάρη στην ε, ε, γεωργία και σε γεωργικές εκτάσεις, γιατί υπάρχουν, υπάρχουν πολύ περισσότερο ελεύθεροι χώροι από ότι στις πόλεις. Υπάρχουν λοιπόν και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της γεωργίας στο κλίμα και υπάρχουν και πάρα πολλές ευκαιρίες. Όσον αφορά τώρα τις γεωργικές τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τη Γεωργία. Νομίζω θα ξέρετε πολλοί από εσά αυτό το σχεδιάγραμμα. Το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ε, οι περισσότερες εκπομπές ε, προέρχονται από την εντερική ζήμωση. Δηλαδή ε, αυτό που αφορά τα ζώα, μιλάμε για το 42 43% εκπομπών του διοικητήτου του άνθρακα από τη γεωργία. Και υπάρχει και κάτι, υπάρχουν και 15% εκπομπές από την αποσύνθεση της κοπριάς. Αυτά από κοινού ε, αντιστοιχούν σε πάνω από 50% των εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα. Ε, το ζωικό κεφάλαιο ε, πολλές φορές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο προφανώς για τις εκπομπές. Οι άνθρωποι επικρίνουν το θέμα του ζωικού κεφαλαίου, αλλά ξεχνάμε ότι περίπου το 30% των εκπομπών έρχονται από το έδαφος, από τον τρόπο καλλιέργειας των εκτάσεων. Ε, άρα δηλαδή και εδώ πρέπει να αναλυφθούν κάποιες δράσεις. Τα στοιχεία που σας αναφέρω εδώ είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως στα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλές εναλλαγές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έχουμε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εκεί το 44% όλων των γεωργικών εκπομπών από αυτές και μόνο τις τρεις χώρες από κοινού. Και ανάμεσα στις χώρες βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικές ε, ε, εναλλαγές. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ότι σε ορισμένους τομείς ε, έχουμε την ε, δέσμευση του διοξιδίου ε, στα βοσκοτόπια. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να περιστούν οι εκπομπές και να καταλήξουμε, μάλλον αυτά που βλέπετε με το πορτοκαλί, είναι το καθαρό επίπεδο εκπομπών. Ε, βεβαίως μπορούμε να εξετάσουμε και τη γεωργία ε, ανατομής, είναι ο πέμπτος τομέας, μεγαλύτερος τομέας, που συμβάλλει στις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Και τα στοιχεία που βλέπετε στη διαφάνεια είναι το επίπεδο των εκπομπών εξαιρουμένων ε, των εκπομπών από τις χρήσεις γης και από τη δασοκομεία. από ε, το πρόγραμμα Λουλούσφ. Υπάρχουν όμως και πολλές εναλλαγές ανάμεσα στις ίδιες χώρες και αυτό που βλέπουμε είναι ότι στο μέλλον η γεωργία θα παίξει όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Αυτή τη διαφάνεια τι βλέπετε από την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Στη μέση της διαφάνειας αυτής βλέπετε τα στοιχεία προς το 2030 και πιο κάτω πάνε μέχρι το 2050. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι το μεγάλο μπλε. Αυτό αφορά τις εκπομπές από τη Γεωργία. Ε, και έχει συμβεί το εξή, έχει συμβεί το εξής. Στους άλλους τομείς έχουν μειωθεί κατά πολύ εκπομπές, άρα δηλαδή το ποσοστό και η συνεισφορά της γεωργίας στις εκπομπές διοικητήτου του άνθρακα αυξάνεται. Κάνοντας μια προβολή στο μέλλον, βλέπουμε ότι η γεωργία ευθύνεται όλο και περισσότερο για την αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Φτάνουμε λοιπόν στο ερώτημα τι θα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το πλαίσιο που ισχύει και τι δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε και πώς ακριβώς μπορούμε να αποκριθούμε στα αιτήματα του, Παρισιού. Τώρα, ε, υπάρχει ένα πλαίσιο αυτό έχει σχέση με το πρωτόκολλο του Κιώτο, ισχύει μέχρι το 2020. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και τη γεωργία. Και όπως ανέφερα προηγουμένως, Εκεί περιλαμβάνονται διάφοροι τρόποι υπολογισμού των εκπομπών ανάμεσα ε, σε που αφορά στους διάφορους τομείς, μεταξύ αυτών ε, και στη γεωργία. Στο πλαίσιο του 2020 υπάρχει επίσης και το ε, πρόγραμμα Λουλούσφ και το πρόγραμμα της δασοπονίας και δασοκομείας το 2030, ε, στις προτάσεις για το 2030 για το πλαίσιο, εκεί θα έχουμε μία αλλαγή. Θα αρχίσουν δηλαδή να συνυπολογίζονται και άλλα στοιχεία, στοιχεία όπου η γεωργία μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Στο πλαίσιο λοιπόν του 2030 βλέπετε το πώς θα εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Παρισιού. Έχουμε το 40% μείωση, ε, στόχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στόχο μέχρι το 2050 να περάσουμε σε 80%. Και φυσικά θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να μειωθούν οι, οι εκπομπές ώστε να φτάσουμε το πολύ σε 1,5 βαθμό αύξηση της θερμοκρασίας, κάτω από το 2 δηλαδή. Τώρα, επίσης έχουμε στη Γεωργία την στρατηγική προσαρμογή στι κλιματικέ αλλαγέ. Κάτι που απαιτεί από τα κράτη-μέλη να ε, ενημερώσουν την Επιτροπή για το πώ αντιμετωπίσουν τι κλιματικέ αλλαγέ. Και η Γεωργία θα παίξει ρόλο κλειδί. Υπάρχουν και άλλε πολιτικέ, ε, υπάρχουσε, ε, η προσαναθεώρηση προκειμένου να εφαρμοστούν οι, κλιμα... οι στρατηγικές για την πολιτική αλλαγή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε ήδη πρόταση για τη Γεωργία θα ακολουθήσει. Τώρα για να δούμε πώς επιμερίζονται οι εκπομπές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της δράσης που θα κληθούμε να λάβουμε. Όπως ανέφερα, οι εκπομπές από Λούλου ΣΥΕΦ ε, έχουν και με διοξίδιο του άνθρακα, από ε, φύτεμα φυτών, από βιομάζα, Επίσης, ε, έχουμε και τον επιμερισμό των προσπαθειών με εκπομπές μεθανίου και οξυδίων του αζότου. Και αυτό είναι, αφορά περισσότερο τη διαχείριση της γεωργικής γης, την ε, εκτροφή σε βοσκοτόπια και τις εκπομπές από τα εδάφη. Κάτι που είναι σημαντικό ενώ των προτάσεων του 2030 είναι η ελαστικότητα μεταξύ των δύο προτινόμενων μηχανισμών υπολογισμού. Ε, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό και τον επιμερισμό των προσπαθειών, προτείνεται κάποιες ε, ε, αφαιρέσει από τον τομέα χρήση γη, αλλαγή χρήση γη και δοσοκομεία να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη για να υλοποιήσουν του δεσμευτικού στόχου σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των προσπαθειών. Και πριν επισέλθω στη συζήτηση αυτών των θεμάτων, θα ήθελα να πω ότι ε, αξίζει να δούμε το επίπεδο εκπομπών των κρατών μελών. Βλέπετε ένα πίνακα με τη με τη μερίδα της ε, γεωργίας ε, σε εκπομπές πλήν του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή με απόβλητα, μεταφορές, ε, κτίρια και γεωργία. Και βλέπετε έχουμε την Ιρλανδία με το υψηλότερο επίπεδο εκπομπών σε ό,τι αφορά τους, την Γεωργία και επίσης Δανία, Λιθουανία και, Λετων... και Λετωνία με υψηλότερες εκπομπές, ενώ η Ιταλία και η Μάλτα είναι στα χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών. Και περνώντας από το 2020 στο 2030 βλέπουμε τους ε, διαφορετικούς στόχους που έχουμε για το 2020 και το 2030 για τα κράτη-μέλη. Βλέπετε ε, τις γκρίζες στήλε και μερικές γκρίζες στήλε άνω της γραμμής ε, που αφορούν το 2030 και λαμβάνονται υπόψη το κατακεφαλήν εισόδημα, ε, ε εμπλεκόμενες χώρες και την ανάγκη να ανταποκριθούμε στους ε, στόχους ε, ε, των κλιματικών αλλαγών. Και ως προς το 2030 οι περισσότερες απαιτήσει αφορούν τις μειώσεις εκπομπών. Δεν επιτρέπεται καμία αύξηση των εκπομπών δηλαδή στα πλαίσια των τομέων ESD, δηλαδή της, του επιμερισμού των προσπαθειών, της οδηγίας για τον επιμερισμό των προσπαθειών. Σε ό,τι αφορά την χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοκομεία, ε, εδώ έχουμε κυρίως λάβει υπόψη το μερίδιο της γεωργίας, γιατί είναι δύσκολο, δεδομένου των πολλαπλών στόχων της γεωργίας που θα πρέπει να διαφυλάξουμε, να υλοποιηθεί. Γι' αυτό και υπάρχει εξέταση του κατά πόσο ο τομέας της γεωργίας στην επιμερισμό των προσπαθειών θα πρέπει να λάβει υπόψη και τον τομέα ε, Λουλουσιεφ, είτε μιλούμε για αναδάσωση, είτε για δέσμευση από τα δάφη, για να περιλάβει και την χρήση γης, αλλαγής χρήσης και δασοκομεία στον επιμερισμό προσπαθειών. Βλέπουμε Λιθωνία, Λετωνία, ε, Ιρλανδία που ανταποκρίνονται στις προσπάθειες επιμερισμού. Βέβαια, ε, ο κανονισμός για τη χρήση γης, αλλαγής, χρήσης γης και δοσοκομεία ε, δεν έχει διπλό κανόνα. Δηλαδή θα πρέπει οι εκπομπές να, αντικατασταθούν από τις ε, αφαιρέσεις. Οπότε αν μια χώρα χρησιμοποιήσει κάποιες ευελιξίες, ο τομέας Λουλουσιέφ θα πρέπει να έχει περισσότερες επιδόσεις ό,τι αφορά την αφαίρεση. Οπότε αυτό ε, καλύπτεται εν μέρη από τον κανονισμό επιμερισμού προσπαθειών, εν μέρη από το Λουλουσιέφ. Το θέμα είναι να βρεθεί μια ισορροπία των εκπομπών. Και πριν δώσω το λόγο στην ε, Κέλλη, θα ήθελα να δούμε ποια θα είναι η συνέπεια για τη γεωργία. Υπάρχουν πολλές πράξεις και ενέργειες μετριασμού και δραστηριότητες ε, που μπορούν να συμβάλλουν στην οποία των κλιματικών στόχων. Μερικές μάλιστα έχουν δοκιμαστεί, είναι διαθέσιμες και καλύπτουν τα βασκοτόπια, τα καλλιεργη... τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, την κτηροτροφία, όπως αλλαγές ε, ε, στην, ε, χρήση της άρρωσης, στη διαχείριση των επιζωτιών και ούτω καθεξής. Αλλά και στο τομέα Λουσιεύ θα μπορούμε είτε να έχουμε νέα αγρο, αγροδασοκομικά μέτρα ή διαφύλαξη των υγροτόπων και τυρφώνων. Νομίζω ότι έτσι θα αυξηθεί η συμβολή και του κλάδο αυτού. Τώρα θα σας μιλήσει συνάδελφος η Κέιλι για την κοινή γεωργική πολιτική. Περνάμε στο δυναμικό της κοινή γεωργικής πολιτικής ό,τι αφορά την προώθηση των κλιματικών δράσεων. Όπως γνωρίζετε, η κοινή γεωργική πολιτική έχει εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου και οι περιβαλλοντικοί της στόχοι έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια και μάλιστα είναι οι ε, περιβαλλοντικοί στόχοι με βάση τη βιώσιμη διαχείριση ε, των ε, φυσικών πόρων και των κλιματικών δράσεων έχει ανακτήσει σημαντική προτεραιότητα, μία από τι τρει σημαντικότερε τη ΚΑΠ, δηλαδή ο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και η προσαρμογή. Οπότε υπάρχει ήδη το πλαίσιο και υπάρχουν μέτρα και μηχανισμοί εντό τη κοινή γεωργική πολιτική που θα επιτρέψουν στην κοινή γεωργική πολιτική να έχει και κάποια περιβαλλοντικά ωφέλη. Και αυτό τονίζεται και στο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει δέσμευση το 20% του συνολικού γεωργικού προϋπολογισμού να αφιερώνεται σε περιβαλλοντικές κλιματικές δράσεις. Και μάλιστα στο έγγραφο εργασίας της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ήδη χρησιμοποίησε το μισό από το ποσοστό αυτό που έχει αφιερωθεί από την ΚΑΠ για τα περιβαλλοντικά μέτρα και χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της ανείχνευσης, αλλά μερικές φορές ήταν υπερβολικός ο υπολογισμός. Υπάρχουν πολλά μέσα λοιπόν και μέτρα που υπάρχουν στην κοινωνική πολιτική και μπορούν να, να καταλήξουν σε περιβαλλοντικές δράσεις, πολλαπλή συμμόρφωση, ε, καλές προδιαγραφές ε, περιβαλλοντικής γεωργίας, ε, αναβίωση των εδαφών. Όλα αυτά συμβάλλουν στη δέσμευση του, του ε, άνθρακα μέσω πυκνής φλάστης, ε, όπως είναι των δασών. Επίσης έχουμε συστήματα με νέα συστήματα πρεσινίσματος στον πρώτο πυλώνα, αλλά και στις δαπάνες για την, για την αγροτική ανάπτυξη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω παροχής συμβουλών για το κλίμα στη Γεωργία. Επίσης έχουμε τις πράσινες άμεσα ε, ενισχύσεις και τις, ε, τα μόνιμα βοσκοτόπια που συμβάλλουν στη δέσμευση του άνθρακα και τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν την, στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Και υπάρχουν και τα μέτρα του πυλώνα 2. Εκεί έχουμε ένα φάσμα μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη διαχείριση της γης των εδαφών, είτε για τις επενδυτικές δραστηριότητες, είτε για τη δημιουργία ικανοτήτων. Και προβλέπεται και σημαντική ευελιξία για τα κράτη-μέλη για το πώς θα εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά. Και μάλιστα ε, στην τελευταία μεταρρύθμιση είχαμε μεγαλύτερη ελαστικότητα και στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Οπότε στην πράξη η υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα που θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και το τι δυνατότητες θα προσφέρουν στους γεωργούς. Αυτό θα επηρεάσει τις δυνατότητες ε, των γεωργών σε τι έχουν πρόσβαση και ποια μέτρα είναι διαθέσιμα. Και φυσικά θα πρέπει να δοθούν ενάυσματα στους γεωργούς να εφαρμόσουν και στην πράξη τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, την παρατηρούμε μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι δεν έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερη φιλοδοξία τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα για περιβαλλοντικούς στόχους διαπιστώνουμε ότι το κλίμα, για παράδειγμα, δεν είναι υποχρεωτικό στοιχείο του συστήματος παροχής συμβουλών στο γεωργό. Και το πρασίνισμα, αυτό το greening, για τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων, δεν εφαρμόζεται παντού. Οπότε, ε, ενώ υπάρχει μια δέσμευση, μετά εκλείεται και πάλι στην ατμόσφαιρα. Ούτε ε, προστατεύονται όλες οι γεωργικές γέες από την άρρωση που θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευθεί αν θα πρέπει, αν θέλουμε να παραμείνει δεσμευμένο στο έδαφος ο, ο άνθρακας. Επίσης, έχουμε διάφορα μέσα, μηχανισμούς και ευελιξία προκειμένου να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών και να τις επιτρέψουμε να υλοποιήσουν τις κλιματικές ε, απαιτήσεις ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αλλά βλέπουμε εδώ από τον πίνακα το σκούρο πράσινο που αφορά την περιβαλλοντική δράση με το βελάκι που δείχνει προς αυτό, που είναι μόνο το 8% του, της προγραμματιζόμενης, της προβλεπόμενης χρηματοδότησης δυστυχώς. Βέβαια, κάποια κονδύλια άλλων κλάδων ίσως έχουν και περιβαλλοντικές συνέπειες, αλλά λέω ότι μόνο το 8% της συνολικής, ε, ε, του συνολικού προϋπολογισμού αφιερώνεται αποκλειστικά στην υλοποίηση περιβαλλοντικών μέτρων. Επίσης, ε, ο τρόπος που γίνεται ο προγραμματισμός και η χρηματοδότηση των επιμέρους προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη επίσης ε, είναι νομιόμορφος. Βλέπετε ε, τις χώρες σε Πορτογαλία που έχουν κάτω από το μέσο όρο εφαρμογή των προγραμμάτων και άλλες πάνω από το μέσο όρο, οι υπόλοιπες. Ε, η Σλοβενία και η Ολλανδία είναι από αυτές που έχουν τις μεγαλύτερες επιδόσεις. Βλέπω ότι πλησιάζουμε στην εξάρτηση του 20 λεπτού. Αν δούμε όμως τους στόχους που υιοθετήθηκαν για το ε, κλίμα στα προγράμματα ανάπτυξης ε, της υπαίθρου βλέπουμε ότι είναι αρκετά χαμηλά τα ποσοστά. Μόνο 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν αφιερωθεί για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση ή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βέβαια, 2,8 δισεκατομμύρια μπορεί να ακούγονται ως υπέρογο ποσό, αλλά είναι λιγότερο από το 2% του συνολικού υπολογισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μόνο 2% των μονάδων κτηνοτροφίας ε, έχουν επενδύσεις για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Και επίσης ε, στα δεξιά βλέπουμε το 1,8% που αφορά τη γη που έχει αφιερωθεί στην δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Χαμηλότερο το ποσοστό το 1,8% γιατί ε, πολλά κρατημέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη χρήση της αγροτικής, της γεωργικής γης ως ε, γη για δέσμευση του άνθρακα. Κάτι που θα τους επιτρέψει να υλοποιήσουν τους περιβαλλοντικούς στόχους. Οπότε έτσι η γεωργία δεν προβαίνει σε σημαντικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, παρόλο που υπάρχει δυνατότητα από τα μέτρα και τους μηχανισμούς της ΚΑΠ. Το δυναμικό υπάρχει, αλλά δεν αξιοποιείται αρκετά. Τέλος, τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα κατάματα για να υλοποιήσουμε τους στόχους που αναλάβαμε και τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε στο Παρίσι. Θα πρέπει να έχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές για όλους τους τομείς ε, γύρω ή μετά το 2050. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ πιο ε, ενδελεχώς το πώς η γεωργία μπορεί να μας βοηθήσει στην υλοποίηση αυτών των στόχων και να διευρύνει το ρόλο της στο μέλλον, γιατί η εκπομπές ε, της γεωργίας θα αυξάνονται σε σχέση με άλλους τομείς. Οπότε θα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ισχυρότερο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η γεωργία, παρόλο που έχει πολυδιάστατο στόχο και έχει ως στόχο την παραγωγή τροφίμων, αλλά ταυτόχρονα έχει ως στόχο την παροχή περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Οπότε η δράση που θα πρέπει να αναλάβουμε θα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ της ε, ανάγκης ανάπτυξης όλων των επιμέρους αυτών στόχων της γεωργίας. Πάντως υπάρχει μεγάλο δυναμικό για ανάληψη δράσης, ε, κάτι που δεν γίνεται αρκετά. Σας ανέφερα προηγουμένως τις δράσεις ε, που μπορούμε να αναλάβουμε, που αφορούν και τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παρά το δυναμικό που υπάρχει, ε, το δυναμικό μετριασμού διαφέρει από δράση σε δράση και από τον τόπο στον οποίο εφαρμόζεται η κάθε δράση. Οπότε, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ε, κάνουμε πολλές συστάσεις στην έκθεση. Καταρχήν χρειαζόμαστε στοιχεία. Θα πρέπει να εντοπίσουμε πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή για να δούμε ποιος, ποιο είναι το δυναμικό μετριασμό των κλιματικών αλλαγών ε, σε, συγκεκριμένε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί δεν έχουμε ακριβώς τα στοιχεία για να προβούμε σε αυτή την ανάλυση. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να θέσουμε σαφέστατους στόχους για τον κλάδο, να διαμορφώσουμε ένα όραμα και, και μια συνεπή πολυδιάστατη προσέγγιση προοδευτική για να υλοποιήσουμε το στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου για ολόκληρο τον κλάδο. Και μάλιστα ο νέος, η νέα πρόταση κανονισμού για τη διακυβέρνηση προτείνει στα κράτη-μέλη να εκπονήσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές πεντηκονταετίες ε, που να περιλαμβάνουν και τη γεωργία και τη χρησιγής αλλά και τη δασοκομεία και θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα θα πρέπει να έχουμε ειδικό στόχο για τη γεωργία στο σύνολό της Και κάτι τέτοιο θα δώσει ενάυσματα στους γεωργούς για να αναλάβουν περισσότερες δράσεις. Ε, και να μην ξεχνούμε και το θέμα της ζήτησης, της κατανάλωσης. Ε, θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση ε, σε προϊόντα που αυξάνουν τις εκπομπές, για παράδειγμα γαλακτοκομικά ή κρέας. Πάντω στην ε, ανέβριση των στόχων θα πρέπει να φροντίσουμε οι πολιτικές που θα εφαρμόσουμε θα είναι σωστές ώστε να έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα εφαρμόζονται με τρόπο ώστε τα μέτρα που είναι διαθέσιμα να εφαρμόζονται και στην πράξη και να μην μένουν μόνο στα χαρτιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση της μελέτης σας. Νομίζω ότι μας λύθηκαν πολλές ε, απορίες, διευκρινίστηκαν πολλά θέματα και θα μπορέσουμε έτσι καλύτερα να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τα θέματα αυτά. Γιατί οι κλιματικές αλλαγές είναι πολύ σημαντικό θέμα και περιέχουν πολλούς κινδύνους, πολλές απειλές, αλλά και σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκαν έχει το λόγο. Ε, thank was, ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Τα τελευταία σας σχόλια θα μου οδηγήσουν σε μια ερώτηση. Είπατε ότι πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός χωστός για να υπάρχουν τα σωστά αποτελέσματα. Εμείς έχουμε στην Ιρλανδία ένα πρόβλημα με το πρόγραμμα για το πρασίνισμα και την χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρωκα. Το πρόβλημα για μας είναι ότι έχουμε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τομέα αυτό και οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς να τους προσελκύσουμε στο να είναι πραγματικά εμπλεκόμενοι και αποτελεσματική σε τέτοιου είδους ε, προγράμματα. Φαίνεται ότι προσπαθούμε με πολύ βαρύκτυπο τρόπο να απλοποιήσουμε κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο περίπλοκο και ουσιαστικά πάρα πολύ αργά απλοποιούμε τον πυλώνα 2. Είναι εύκολο να κατηγορεί βέβαια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως εδώ η αλυσίδα λήψη αποφάσεων είναι πάρα πολύ αργή. Στην πράξη δεν βλέπω λοιπόν να προχωρεί το πρόγραμμα αυτό. Ακούσαμε πολλούς να μιλούν για την κλιματική αλλαγή, για την πολιτική και για τον συμπληρωματικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την πρόταση που ακούσαμε, θα πρέπει να στέλνουμε βόλιο κρέας υπερατλαντικά και προϊόντα ε, από την Αμερική. Τι να ε, εισάγουμε, τον ρωτήσαμε και μας απάντησε αμύγδαλα. Κοιτάξτε, ε, για μένα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι προσπαθεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό και δημιουργούνται και πάρα πολλά ερωτήματα. Δύο λεπτά και όχι δευτερόλεπτο, ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Άγνιο. Πριν από 31 χρόνια ε, στην Αγγλία ε, είχα παρακολουθήσει μία διάλεξη για την ε, υπερθέρμανση του πλανήτη. Και εκεί είχαμε του επιστήμονε, γιατί μου λέγανε, που έλεγαν ότι μετά από 30 χρόνια, πέρυσι δηλαδή ήταν η τελευταία χρονιά, πρόκειτο να βιώσουμε τελείω διαφορετικό κλίμα με πιο ζεστούς χειμώνε και πιο ξερά καλοκαίρια. Θα αυξανόταν γινόταν η στάθμη του υδάτων, αλλά δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά τραγικά. Και νομίζω, εγώ ξεκίνησα το 1971 τότε ε, τη Γεωργία, πριν από έξι χρόνια είχαμε τον πιο σκληρό χειμώνα, ε, τότε πραγματικά πάγωσαν τα πάντα. Ακόμα και πέρυσι είχαμε βροχερό καλοκαίρι, έτσι πρέπει να τα δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η Συμφωνία του Παρισιού δεν λέει ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι πιο σημαντική και από το να πρέπει να ε, βελτιώσουμε τον καιρό ε, στον κόσμο. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να λάβει μέτρα και στόχους για τα κράτη-μέλη. Προφανώς ε, η Γεωργία εκπέμπει. Χρειαζόμαστε όμως να υπάρχουν λιγότερες εκπομπές εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι τουλάχιστον αυτό εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τα οξύδια αζότου ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί αν ε, τα ε, περιορίσουμε σημαίνει ότι θα έχουμε και μικρότερες εκτινοτροφικές μονάδες. Μπορεί μερικοί να μπορούν να το δεχτούν αυτό, όχι όμως η Ιρλανδία και αυτά αφορά και εσά. και η δική σας εκτινοτροφία θα υπάρχει υποστεί ζημιές. Γι' αυτό λοιπόν ε, βεβαίως και θα εισάγουμε τη διαφορά. Ίσως το 20% να αφορά τις ε, πληρωμές αυτές που εκκρεμούν για τους γεωργούς ε, ας μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει ο κίνδυνος των πυκαγιών και από εκεί εκπομπές του ε, διοξιδίου του άνθρακα. Στην ίχνη λασιμότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους γεωργούς. Εν μεταξύ υπάρχει υποκρισία ότι ε, για, τους, για την νερό διαχώνευση καλλιεργείται το καλαμπόκι και αυτό δεν ισχύει. Σε τελική ανάλυση, αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί να προσπαθούμε να ασχολούμεθα με όλα. Σας ευχαριστώ. Ε, ίσως ε, δεν ε, κάνετε τη συγκομιδή των ζαχαρότευτων εγκαίρος, γι' αυτό σας πάγωσαν. Ο κύριος Λαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ε, οργανώσεις ε, γεωργών θεωρούν ότι θα αυξηθεί η κερδοσκοπία μετά την COP21. Αυτή η COP21 είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των ε, καλλιεργήσιμων ε, περιοχών, της ε, αποψήλωσης και πολλών από τον κακό που αντιμετωπίζουμε. Και βεβαίως η αλλαγή του κλίματος έχει επιπτώσεις στη γεωργία. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για την αμπελουργία. Πριν από πολλά χρόνια βλέπαμε οι εποχές να διαρκούν πάνω από δύο μήνες με σταφύλια πολύ πιο όρημα, πιο γρήγορα και πιο γλυκά. Αυτό είχε επιπτώσεις στην καλλιέργεια των αμπελιών εδώ και πολλά χρόνια. Έχει αυξηθεί σιγά σιγά η θερμοκρασία κοντά στην περιοχή του Λίγυρα. Το ίδιο και στην Μεγάλη Βρετανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ότι σημαντικά έχει αυξηθεί η παραγωγή των αμπελιών χάρη σε αυτήν την αύξηση της θερμοκρασίας και πολλές παραγωγές είτε εξαφανίζονται είτε αυξάνονται. Βλέπουμε λοιπόν την ευρωπαϊκή πολιτική η οποία δεν προσαρμόζεται σε αυτά τα δεδομένα και όλες οι χώρες δεν μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Οι άλλες χώρες τι έχουν κάνει. Δεν θα ήταν ορθό κάποιες χώρες να ακολουθούν αυτούς τους πολύ αυστηρούς κανόνες, ενώ άλλες τους αγνοούν. Κυρία Σλάιερ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση της μελέτης, γιατί άκουσα πολλά θετικά στοιχεία και πολλές ευκαιρίες που διανοίγονται. Γιατί είπατε ότι μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε υγιή τα εδάφη μας και έχουμε και γι' αυτό και την οδηγία πλαίσιο για το νερό. Και φαίνεται ότι τάσσεστε υπέρ τη περιφερειοποίησης, ώστε να αναλαμβάνει και ο Γιώργος την ευθύνη. Είστε υπέρ της έρευνας, της καινοτομίας, της ανακύκλωσης των ε, οργανικών ουσιών, αλλά είστε και πέρα της πιο περιορισμένης χρήσης των λοιπασμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε οι δύο επιτροπές γεωργίας και περιβάλλοντος. Και επίσης, ας μην ξεχνούμε ότι στην Ολλανδία ήταν καταστροφική η εφαρμογή της οδηγίας για τα ζωτούχα λοιπάσματα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σίγουρα η κατάσταση επιτόπου, ξεκινώντας από την ε, ανάγκη ότι χρειαζόμαστε ποιοτικά εδάφη και ποιοτικό νερό. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι μας ενδιαφέρουν και βιώσιμες ε, θέσεις απασχόλησης. Ο κύριος Κάρθη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλλαγή του κλίματος βεβαίως και επηρεάζει πολλές περιοχές, αλλά κάποιοι βρίσκονται πολύ μακριά από την κλιματική αλλαγή είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα μπορούν να διαπιστώσουν ότι υπάρχει, ότι είναι μια απειλή για την ύπαρξή τους. Και αναφέρομαι εδώ στους ε, γεωργούς οι οποίοι οργώνουν στη δική μου εκλογική επικράτεια και στην περιοχή μου βλέπουμε ότι σαφώς αυτές οι πολύ σκληρές ε, κλιματολογικές συνθήκες τους έχουν επηρεάσει. Και πραγματικά οι περισσότεροι από αυτούς τους γεωργούς θέλουν να παίξουν ένα ρόλο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Το πρόβλημα είναι όμως ότι στις περισσότερες περιπτώσεις παίρνουν πολύ αντιφατικά μηνύματα για το τι πρέπει να κάνουν. Ξέρω ότι κάποιοι θα πούν ότι δεν πρέπει να τρώμε καθόλου παραδείγμα παραδείγματος χάρη. Όμως πολλοί χαίρονται και τους αρέσει να τρώνε από καιρούς καιρών βοηοκρέας. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκτρέφουν τα ζώα χρειάζονται βοσκοτόπια, χρειάζονται χορτάρι. Και εκεί ξεκινάει αν θέλετε και η αντίφαση με τους στόχους που έχουμε υιοθετήσει και με τις ανώτατες τιμές για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει μια αναγνώριση ότι εδώ έχουμε υιοθετήσει αντιφατικούς στόχους. Και δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια, αλλά υπάρχει αντίφαση απόλυτη αντίφαση. Από τη μία υιοθετούμε πολιτική για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, από την άλλη έχουμε τους στόχους για το βόλιο κρέας, έχουμε τις εμπορικές συναλλαγές και τις συμφωνίες που αφορούν το εμπόριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ανησυχούν οι γεωργοί μας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Έχετε άποψη όσον αφορά την εξάλληψη αυτών των αντιφάσεων, διότι καταλαβαίνετε ότι οι γεωργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτές τις αερολογίες και πολλές φορές δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε και εμείς τι να τους πούμε ε, ότι είναι η σωστή κατεύθυνση. Ο ε, ε, Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους εισηγητές για την πάρα πολύ καλή εισήγησή τους, μια πάρα πολύ καλή μελέτη, η οποία είναι και πολύ χρήσιμη για μας. Εγώ ε, παρεμβαίνω ως ε, εισηγητής της Επιτροπής Γεργίας σχετικά με αυτόν τον κανονισμό effort sharing, ε, τον επιμερισμό των προσπαθειών. Τον αναφέρετε και εσείς ε, στην εισηγησή σα. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και εδώ και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ο μετριασμός. Στη σελίδα 10 της μελέτης σας αναφέρεται ότι είναι αδιαμφισβήτητο. Υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη παραδοχή. Με βάση αυτή Όσο πιο δαπανηρό είναι η παραγωγή στη Γεωργία, όσο πιο δαπανηρή είναι η Γεωργία, αυτό μετακυλείται και σε άλλου τομεί, παραδείγματο χάρη στι μεταφορέ. Μήπω μπορείτε να μα δώσετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για να μα εξηγήσετε πού βασίζεται αυτή την υπόθεσή σα. Και ξεκινώντα από αυτό, εσεί πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο η ευελιξία Λουλουσιέφ ε, που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών να ε, διαπιστωθεί πόσο σημαντικό είναι να σκεφτούμε πιο κατάλληλες ε, δυνατότητες έτσι ώστε και ο ίδιος ο τομέας να συμβάλλει στο μετριασμό και στη δέσμευση των αερίων του θερμοκηπίου κυρίως μέσα από την εφαρμογή του ε, κανονισμού LULUCF. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η γεωργική πολιτική και η προστασία του περιβάλλοντος εκπέμπουν μηνύματα που είναι αντιφατικά. Το είπε και ο προλαλής σας και θα ήθελα να σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Ίσως μπορείτε να τοποθετηθείτε από αυτόν. Το πρώτο παράδειγμα ε, έχουμε όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θέλουμε να περιορίσουμε τα απόβλητα ε, και θα μπορούσε κανείς ε, να ε, υποθέσει ότι με τον τρόπο αυτό αποδεσμεύονται γεωργικές εκτάσεις. Ναι, αλλά αν εκεί χρησιμοποιούνται δίζελ και άλλου τέτοιου είδους καύσιμα, εσείς τι λέτε, αυτό είναι καλό, επειδή δεν θα ε, χρειάζεται να εισάγουμε πετρέλαιο. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτόν τον τομέα βασίζουμε σε λάθος κατεύθυνση. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε ε, την χρήση ε, των λοιπασμάτων όπου δεν χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν άλλες όπου δεν χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους λοιπάσματα. Αν λοιπόν δεν επιτρέπεται η χρήση λοιπασμάτων, δεν θα υπάρχουν και πια κάποιες καλλιέργειες. Σε αυτές τις 300.000 εκτάρια θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε μεταξύ άλλων σόγια, δηλαδή 45 εκατομμύρια δίζελ για τις μεταφορές επιπρόσθετα. Και αυτό όμως είναι ένα αντιφατικό μήνυμα, γιατί δεν θέλουμε να καλλιεργούμε φασόλια και μπιζέλια, τα εισάγουμε και τι γίνεται, αυτό δεν είναι καλό για την προστασία του κλίματος. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα έπρεπε άραγε στην γεωργική πολιτική να εκπέμπουμε ε, μη αντιφατικά μηνύματα. Γιατί αυτό που είναι απαραίτητο να υπάρχει είναι μια αξιόπιστη και σταθερή γεωργική πολιτική. Εδώ δεν πρόκειται για τα χρήματα, ε, πρόκειται για τη στρατηγική να μπορεί ένας επιχειρηματίας να προσαρμοστεί σε μια, σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. παρακαλώ. Ναι, νομίζω ότι η μη χρησιμοποίηση παραστοκτώνων και αν μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε το παράδειγμα άλλων των βιολογικών ε, αγροκτημάτων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θα ήθελα όμως να κάνω την εξή ερώτηση. Εδώ υπάρχουν βεβαίως επιστήμονες που πρεσβεύουν τη μία ή την άλλη άποψη και δεν συμφωνούν. Το θέμα της μεθόδου χωρίς άρρωση και αν αυτή είναι η πιο αποτελεσματική. Ξέρετε ότι αυτό επίσης αμφισβητείται στο Ινστιτούτο στην Γερμανία λέει ότι δεν είναι μέτωπο που προστατεύει από την κλιματική αλλαγή και δεν το ζητούν πλέον τα περισσότερα από τα γερμανικά κρατήδια. Υπάρχουν όμως άλλες μελέτες που λένε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το μέτρο με την προστασία από την αλλαγή του κλίματος. Και όσον αφορά το ηλαρό αέριο, και εδώ υπάρχουν διαφορετικές επιστημονικές ε, μελέτες και απόψεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο κατώτατο όριο, στα όρια όπως έχουν θεσπιθεί και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι γεωργοί εδώ να δουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σύνδεση με την γλυφοσάτη, γιατί και εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης. Πάντα με ξαφνιάζει το θέμα της χρήσης ή όχι αυτών των ουσιών. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της χημικής βιομηχανίας και το θέμα του, των εκπομπών αζότου, διοξιδίου του άνθρακα και αυτό είναι κάτι που επιβαρύνει το περιβάλλον και ο γεωργός θα πρέπει να είναι φιλικός προς το περιβάλλον, να χρησιμοποιεί βιώσιμα συστήματα και να αποφεύγει αυτά που μολύνουν το περιβάλλον, καθώς και την ε, εντατική, κάθε είδους εντατική εκμετάλλευση και καλλιέργεια. Αυτά. Ο κύριος Ροπέ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτής της ενδιαφέρουσας μελέτης και τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που δώσατε και που θα αξιοποιηθούν όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα κράτη-μέλη. Γιατί θα δουν με τους πίνακες σε τι θέση βρίσκονται και μπορούν να λάβουν δράσεις για να βελτιώσουν την κατάσταση. Αν κατάλαβα καλά, σε πολλές χώρες όπως τη Λιθουανία υπάρχει τελείως εγκαταλελειμμένη υγεία, χρησιμοποίητη. 5% των εδαφών στη Λιθουανία είναι γη ανεκμετάλλευτη. Οι ιδιοκτήτες δεν ξέρουν πώς να την χρησιμοποιήσουν, πώς να την αξιοποιήσουν. Και μέσα σε λίγα χρόνια γεμίζουν με ζυζάνια και με χορτάρι. Υπάρχουν όμως φορείς που ελέγχουν αυτούς τους ιδιοκτήτες και τους υποχρεώνουν να ξεχερσώσουν τα χωράφια τους και να αποκαταστήσουν συνθήκες βέλτιστης γεωργικής πρακτικής. Ερωτώ λοιπόν, χρειάζεται εδώ αυτή η περιβαλλοντική δράση, γιατί μερικές φορές ακόμη και ε, ε, αναξιοποίητη η γη είναι χρήσιμη για το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται σαν και καλά να καλλιεργούμε τα πάντα. Κυρία Σκότ Κάτω, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα καταλάβετε και την πληροφορά μου, είμαι Βρετανίδα και εμείς ε, αντιμετωπίζουμε πολύ, με πολύ διαφορετικό τρόπο πια τη γεωργική πολιτική. Γι' αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να σκεφτώ πώς θα εξελισσόταν η, Ευρωπα... γεωργική πολιτική αν δεν περιοριζόταν από την κοινή γεωργική πολιτική. Είμαστε αρκετά επικριτικοί ε, και στην ΚΑΠ αλλά και στο Greening, οπότε άφησα την φαντασία μου να οριάζει προς αυτήν την κατεύθυνση τώρα, στο βρετανικό πλαίσιο εννοείται. Πάντως ε, πολύ χρήσιμη η μελέτη και σχετική ακρόαση, γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε τη Συμφωνία των Παρισίων, είδαμε ότι ο κλάδος γενικώ έλαβε το μήνυμα για τη σημασία που έχει ο μετριασμός των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση των ορεικτών καυσίμων και θα πρέπει στο μέλλον η βιομηχανία να αρχίσει να δρά με διαφορετικό τρόπο. Εθαρρυντικά όλα αυτά. Αλλά οι κλιματικές αλλαγές έχουν φτάσει ήδη σε υψηλά επίπεδα. Βλέπετε πώς λιώνουν οι παγετώνες ε, στην Αρκτική. Και θα πρέπει να απορροφήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα που ήδη είναι ελεύθερο στην ατμόσφαιρα και σίγουρα η σωστή διαχείριση της γης είναι ένας τρόπος για να το επιτύχουμε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά την αλλαγή της διατροφής, τι γνώμη έχετε. Εμείς στην, στο κόμμα μου είμαστε υπέρ της μεταστροφής προς μια φυτοφαγική διατροφή. Δεν έχω εστεριστεί πλήρως αυτή την ε, φυτοφαγία, αλλά το σκεφτόμαστε. Ποια λοιπόν θα είναι μια βιώσιμη γεωργία στο βρετανικό πλαίσιο. Ε, σκεφτόμενοι αυτό, είπαμε να προσθεθεί η περιεκτικότητα ε, του λίπου στο κρέας για να το χρησιμοποιήσουμε, να το προσαρμόσουμε ως, ε, ως προϊόν πολυτελείας. Επίσης, για να στηρίξουμε το βιοπορισμό των γεωργών. Αν γίνει με μεταστροφή σε μια φυτοφαγική διατροφή ε, των καταναλωτών ε, και αν ο κόσμος αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά τη γεωργία, θα πρέπει ταυτόχρονα να στηρίξουμε και τους γεωργούς για να προσαρμοστούν σε αυτή τη μεταστροφή. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του εδάφους, δεν είδα και πολλές λεπτομέρειες στη μελέτη σας για αυτό το θέμα. Ένα ζωντανό έδαφος μπορεί να συγκρατήσει πολύ περισσότερο τον άνθρακα, γιατί βακτηρίδια που χρησιμοποιούν το μεθάνιο θα περιορίσουν και τις ε, εκπομπές σε μεθάνιο από την εντερική ζήμωση των αγελάδων. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Στα συμπεράσματά σας διαπίστωσα ότι μιλάτε και για έλλειψη στόχους όσον αφορά τη γεωργία και την αλλαγή του κλίματος. Και αυτό το βλέπω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είμαι εδώ και δύο χρόνια μέλος αυτής της Επιτροπής και διαπιστώνω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ε, έχουμε προτάσεις που να προέρχονται από τους ίδιους τους γεωργούς. Δεν δεσμεύονται δηλαδή και δεν συμμετέχουν αρκετά στη διαδικασία και με επιμονή θα έλεγα ότι η Γεωργία είναι μια ειδική περίπτωση. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό ότι η Γεωργία θα μπορούσε να είναι ένα διαφορετικό θέμα, ένα ξεχωριστό θέμα. Ε, συμφωνείτε σε αυτό ή το αρνείστε. Και δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να σας κάνω. Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, λίγο πιο συγκεκριμένοι στις πρακτικές συστάσεις ε, που κάνετε. Γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δράσουμε και να σταματήσουμε να μιλάμε. Ο κύριος Ανδρίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές για την παρουσίασή τους. Συμφωνώ σε πολλά από αυτά που μας παρουσιάζουν. Τελικά βλέπουμε ότι υπάρχει το ερώτημα για την κότα και το αυγό. Το κλίμα επηρεάζει τη γεωργία. Η γεωργία επίσης επηρεάζει το κλίμα σήμερα. Και αυτό είναι σωστό, η αλλαγή του κλίματος. Σίγουρα, αυτό το ακούσαμε από πολλούς ομιλητές, οδηγούν ε, σε διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας και γεωργίας τα πράγματα εξελίσσονται ταχύτητα και αν κοιτάξουμε όσον αφορά την COP21 και το πρόβλημα του κλίματος, δεν μπορεί η Γεωργία να παραμείνει εκτός ε, καθότι δεν είναι ο μόνος ε, υπέτειος, αλλά σίγουρα βάσει των πορισμάτων που έχουμε σήμερα επηρεάζει και η γεωργία. Η αλλαγή λοιπόν της μεθοδολογίας, της καλλιέργειας. Μιλήσαμε για την κτηνοτροφία, παραδείγματος χάρη και το βόλιο κρέας. Η αλλαγή, αν θέλετε, της ε, επιλογής τροφίμων, αλλά και των ζωοτροφών, θα μπορούσε σιγά σιγά, δεν πρόκειται να αλλάξουμε από τη μία μέρα στην άλλη τρόπους καλλιέργειας και παραγωγής, γιατί αλλιώ ο αγροτικός κόσμος δεν θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει, αλλά οι τρόποι γεωργίας, καλλιέργειας, παραγωγής θα πρέπει σίγουρα να συνεισφέρουν στην μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Βλέπουμε σήμερα ότι σίγουρα η γεωργία θα πρέπει να παίξει το ρόλο της. Το ίδιο όμως και οι μεταφορές και ο τουρισμός και η κατασκευή, η δασοκομεία, η χρήση της γης και να γίνει ένας υπολογισμός των εκπομπών. Έχουμε σήμερα κάποιες, κάποια μοντέλα που βασίζονται σε προσωμιώσεις. Ο τρόπος εκμετάλλευσης της γης και οι άλλοι τρόποι παραγωγής και καλλιέργειας θα πρέπει να εκτιμηθούν σωστά έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλες αυτές τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα παρακαλέσω τους καλεσμένους μας να σχολιάσουν αυτά που άκουσαν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ένα τεταρτάκι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ήταν ε, πάρα πολύ επί της ουσίας. Ε, θα ήθελα να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερες μπορώ και μετά θα δώσω το ρόλο στον Μπεν. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα από τα θέματα που τέθη αρκετά από αρκετούς από εσά ήταν αυτό το θέμα ε, της γεωργίας ως τομέα και κατά πόσον ε, και πώς ε, πρέπει η γεωργία να χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων. Ε, ποιος είναι ο ρόλος της γεωργίας και σε σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος του κλίματος. Ένα πράγμα θέλω να πω, ότι νομίζω θα πρέπει λιγάκι να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Το πώς αντιμετωπίζουμε τη γεωργία γενικότερο στο τομέα και πώς η γεωργία ε, βρίσκεται και σε σχέση με τις ε, περιβαλλοντικές μας προτεραιότητες. Γιατί πολλά από αυτά που προτάθηκαν, που θα ωφελήσουν ε, το κλιματικό πρόβλημα, θα ήταν όμως ωφέλιμα και για τη γεωργία, για την καλλιέργεια των εκτάσεων. Ε, μακροπρόθεσμα ε, θα υπήρχε μεγαλύτερη αντοχή ε, και από πλευράς περιβαλλοντικής και οικονομικής. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και όταν μιλάμε για τη γεωργία, πολύ συχνά μιλάμε και για εκπομπές που δεν είναι διοξίδι του άνθρακα, για μεθάνιο, παραδείγματο χάρη, που είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκπομπέ. Όμω τη Γεωργία πρέπει να αντιμετωπίζουμε σαν ένα σύνολο και είναι ένα από τους λίγους ε, τομεί όπου πράγματι μπορεί να αφαιρεθεί το διοξίδιο από την ατμόσφαιρα. Ετέθη το ερώτημα μήπως θα πρέπει ε, να επεκτείνουμε την ευελιξία με το LULUCF και τις προτάσεις που υπάρχουν για να επιτύχουμε τους στόχους του μετριασμού. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τελική ανάλυση αυτή η απόφαση για την ευελιξία έχει σχέση με το πώς θα προχωρήσουμε, δηλαδή πώς ακριβώς θα προσπαθήσουμε να αναλάβουμε δράση στον τομέα, στο σύνολό του. Και αυτό που έχει σημασία είναι ακριβώς αυτό ότι δεν μπορούμε ε, να δρανούμε. Ο γεωργικός τομέας πρέπει να λάβει δράση ή ένας πολύ ιδιαίτερος τομέας με την έννοια ότι έχει να φτάσει πολλούς στόχους σε την παραγωγή τροφίμων όπως και μία σειρά άλλων στόχων αλλά αν δεν αρχίσουμε να κάνουμε κάτι τώρα τότε στο μέλλον θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο πόνος, οι οδύνες, γιατί το 30, το 20-30 ε, θα πρέπει να λάβουμε περισσότερα μέτρα αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας το 2050 που είναι μηδενικές εκπομπές. Αυτό είναι σημαντικό τώρα να βρεθούν οι λύσεις από το να περιμένουμε τα 20 χρόνια για να μεταφέρουμε τα... τις αποφάσεις, κάτι όμως που θα καταστεί αναπόφευκτο. Υπήρξε και ένα συγκεκριμένο σχόλιο ε, σχετικά με τα παρασιτοκτόνα ε, εγώ εργάζομαι πολύ για τα μέτρα πρασινίσματος ε, στην αγορά. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι οι EFA, οι περιοχές που είναι σχεδιασμένες βιολογικά, ecologically focused areas, αυτές, σε αυτές τις περιοχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται λιπάσματα και ζυζανιοκτώνα στην περίπτωση αυτή σίγουρα θα μειωθεί η παραγωγή. Όμως αυτές οι οικολογικές περιοχές είναι το 50% της, ε, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ε, κατόπιν τούτου ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου κατά πόσον θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση των ζυζανιοκτώνων σε αυτές τις περιοχές. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω, σχετικά με την ε, μηδενική άρρωση. Αυτό ε, θα το κοιτάξω, θα το ελέγξω ε, και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες πράξεις μετριασμού οι οποίες μπορούν να είναι εποφελείς, αποφέρουν δηλαδή ωφέλη μόνο σε κάποιες συγκεκριμένε κλιματικές ζώνες. Ε, το να μειωθεί, να μηδενηθεί το όργωμα, αυτό αξίζει σε άνυδρες περιοχές, ε, παραδείγματος χάνει στη Μεσόγειο. Εκεί είναι αποτελεσματικές, αλλά λιγότερο ε, αποτελεσματικές σε, πιο, σε διαφορετικά κλίματα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να δούμε πού να εφαρμόζουμε ποιες πράξεις, ποιες ενέργειες. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι λεπτομερέστερες μελέτες για τα τεχνικά στοιχεία, για την επιστήμη που μπορεί να στηρίξει, έτσι ώστε να προκύψει πραγματικά μια διαφορά. Διότι η επιστήμη εξελίσσεται προφανώς ε, και ως εκ τούτου πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το δυναμικό μετριασμού που μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορα ε, μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο παντού και αυτό έχει σημασία. Μπεν, θα ήθελες απαντήσεις εσύ στα υπόλοιπα. Ναι, ευχαριστώ Κέλλη. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα το στο θέμα της γεωργίας και το πώς μπορεί να επηρεάσει. Αν και αν ο Γιώργος είναι ειδική περίπτωση αν θέλουμε να επηρεάσουμε τις δράσεις στη Γεωργία, θα πρέπει να επηρεάσουμε 10 και 10 εκατομμύρια γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε ε, για να πειράσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία και να επικεντρωθούμε σε 25 βασικές, βασικά εργοστάσια. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο από αυτή την άποψη να δράσουμε σε άλλους τομείς όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι λιγότεροι από ό,τι στη Γεωργία που είναι 10 εκατομμύρια και. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να επηρεάσουμε την γεωργία και υπάρχουν ευκαιρίε ε, ώστε να προκαλέσουμε την αντίδραση των γεωργών και προσπαθούν να ανταποκριθούν και οι γεωργοί γιατί επηρεάζονται από τι κλιματικέ αλλαγέ και θα πρέπει να του εφοδιάσουμε τα εργαλεία για να μπορέσουν να προσαρμοστούν, να μειώσουν τι ε, εκπομπέ ε, αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι θετικό. Τώρα είναι πιο δαπανηρή μια τέτοια προσπάθεια. Εξαιρετική ερώτηση και μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ε, εξετάσουμε από πού προέρχεται κάτι τέτοιο. Αναφέρεται τη σελίδα 10 της έκθεσης. Ε, βέβαια, φαίνεται ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικό και πολύ πιο δαπανηρό να έχουμε μετριασμό των κλιματικών αλλαγών χάρη σε επεμβάσει στη γεωργία από ό,τι σε άλλους τομείς. Βέβαια, ως ερευνητής θα ήθελα να πω ότι η απάντηση που λαμβάνουμε από το δυναμικό της γεωργίας για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου εξαρτάται από το πώ αντιμετωπίζουμε το κόστος μετριασμού του κλάδου, αν κρίνουμε ότι είναι πιο δαπανηρό ή όχι, ε, τι τίμημα βάζουμε σε διάφορες δραστηριότητες. Πολλά μπορούν να γίνουν και στη γεωργία, πολύ περισσότερα και αυτό φάνηκε και από, τη μελέτη επιπτώσεων ε, και από τον κανονισμό για τον επιμερισμό προσπαθειών και για το τμήμα χρήση γη, ε, αλλαγή χρήση γη και τασοκομεία. Και με χαμηλής, ε, χαμηλού τιμήματο ε, σχετικά ολιγοδάπανε μεθόδου μπορούμε να μετριώσουμε κατά 8% της μειώσει εκπομπών από τον τομέα με βάση τα μοντέλα που έχουμε χρησιμοποιήσει και τις προβλέψεις που έχουμε κάνει. Αλλά ε, παραλαμβάνω, πρέπει να επηρεάσουμε 10 εκατομμύρια και γεωργούς και για να κάνουμε κάτι τέτοιο χρειάζονται προσπάθειες, χρειάζονται πολλές στοχευμένες λύσεις για συγκεκριμένες χώρες, ε, λαμβάνοντα ε, υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών. Επίσης έχουμε επιμέρους κλάδους στη γεωργία, κτηνοτροφία, γαλακτοπαραγωγή και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες στον κλάδο και δεν είναι πολύ δαπανηρή η δράση τώρα. Θα είναι πολύ πιο δαπανηρή αν περιμένουμε και αναβάλουμε τις δράσεις για το μέλλον. Επίσης, ε, δεν θα πληρώσει την ύφη μόνο η κτηνοτροφία. Πολύ συχνά όταν έχουμε τέτοια, τέτοιες συζητήσεις, μην ξεχνάτε ότι 38% ε, των εκπομπών προερχόνται από τα εδάφη, από τη γεωργία δηλαδή. Οπότε αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές του κλάδου θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στα εδάφη, όχι μόνο στην κτηνοτροφία. Οπότε χρειαζόμαστε μια ευρεία φάση σε όλους τους τομείς ε, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σε ό,τι αφορά τα θετικά στοιχεία, φυσικά είναι πρόκληση η μείωση των εκπομπών. Και ε, η γεωργία κτηνοτροφία υστερεί σε σχέση με του άλλου τομεί ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν είναι ανέφικτο κάτι τέτοιο ούτε υπερβολικά δαπανηρό. Και εκεί έχουμε τα θετικά στοιχεία. Οι χρήστε γη, ιδιαίτερα στη γεωργία, μπορούν να διαδραματίσουν κέριο ρόλο ηγετικό και να πρωτοστατήσουν στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, βοηθώντα και άλλου τομεί. Μπορεί να πρωτοστατήσει λοιπόν ο κλάδο στο μετριασμό και να προχωρήσει και από ότι να αντιμετωπίζεται ως ο κλάδος που είναι ο χειρότερος μαθητής και ότι πρέπει ακόμη να εντείνει τις προσπάθειες και να μειώσει εκπομπές. Πριν ξαναδώσω το λόγο στην Κέλλη, θα ήθελα να πω ότι είχαμε πολλά σχόλια για τις εισαγωγές. μερικά πράγματα εισάγουμε, άλλα προϊόντα τα εξάγουμε. Εγώ δεν είμαι ε, εμπειρογνώμονας για τα θέματα του εμπορίου, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά υπάρχει η συνέπεια της διαρροής, ε, της συνέπειας των ε, προσπαθειών μετριασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εμείς θέλουμε, ας πούμε, να μειώσουμε την παραγωγή και έτσι να μετριάσουμε τις εκπομπές μας ή να περιορίσουμε τις δράσεις μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σταθερή ζήτηση ε, τροφίμων. Αν όμως ε, μειώσουμε εμείς τις προσπάθειές μας, θα αναγκαστούμε να εισάγουμε από άλλες, από τρίτες χώρες. Και άσχετα από το τι πιστεύει κανείς, βλέπει τη διαφορά, ό,τι και αν εισάγουμε αμύγδαλα ή κρέας. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το δυναμικό μετριασμού του κάθε κλάδου και να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτό. Και πολύ σωστά αυτό που είπε ο κύριος ε, Κέλλη για, την κατανάλωση. Γιατί θα πρέπει να το δούμε όχι μόνο ως καταναλωτές ή από τη σκοπιά της Γεωργίας, αλλά και από τη σκοπιά του εμπορίου, ώστε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Η Κέλλη πάλι. Ένα τελικό σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο που άκουσα, νομίζω δεν απάντησα σε αυτό, που αφορά πώς ε, θα μπορέσουμε να εμπλακούν και οι γεωργοί σε αυτή τη δράση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο τι ακριβώς αποτέλεσμα έχουμε, αλλά ποιο τρόπο επιλέγουμε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και βεβαίως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το τι γίνεται στην πράξη. Εάν προβλέψουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάποιων πολιτικών αποφάσεων μιας πολιτικής, τότε ενδεχομένως θα υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ του γεωργού, του αγρότη και αυτών που τελικά είναι οι αρμόδιες αρχές. Πιστεύω λοιπόν ότι αν υπάρχουν πολύ αυστηροί έλεγχοι και προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα τα οποία δαπανώνται, δαπανώνται για το σωστό αποτέλεσμα και με το σωστό τρόπο πρόκειται για δημόσια κονδύλια, των οποίων ε, η χρήση πρέπει να είναι αυτή για την οποία έχει ληφθεί απόφαση. Όμως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οδηγήσουμε τους αγρότες σε μια απομάκρυνση, σε μια έλλειψη κινήτρων και μια αποθάριση, απογοήτευση. Οι πληρωμές είναι ένα θέμα και νομίζω ότι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει, πρέπει να μάθει να το ελέγχει. Αλλά το θέμα του επίπεδου των ποσών που καταβάλλονται, το θέμα των κινήτρων, πώς σχεδιάζονται αυτές οι πληρωμές ακριβώς. Και όσο προχωράμε στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών, πιστεύω ότι πολλά από αυτά που ακούστηκαν εδώ είναι ότι ναι, υπάρχει η εργαλειοθήκη, γιατί δεν λειτουργεί, γιατί στην πράξη δεν φαίνει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Οι γεωργοί πολλές φορές βλέπουμε να μην συμμετέχουν. Πολλές φορές φταίνε τα κράτη-μέλη που δεν είναι διατεθειμένα ή δεν χρησιμοποιούν τη σωστή μέθοδο εφαρμογής. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι η έλλειψη αποτελεσμάτων οφείλεται στη μη συμμετοχή των ίδιων των γεωργών. Μάλιστα. Εξαντλήσαμε και το χρόνο της απάντησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους μας γιατί ήταν πολύ αξιόλογη, άρτια και μεστή μελέτη και η παρουσίαση επίσης πολύ διαφωτιστική και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία, τη συνεργασία μας. Θα αξιοποιήσουμε και τη μελέτη σας και φαντάζομαι ότι θα ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η παρουσίαση. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Έχει έρθει ο κύριος Τιμπορσάνη, ο εισηγητής της γνωμοδότησης. Είναι το τελευταίο σημείο της απογευματινής ημέρησης διάταξης και αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό του 2018. Όπως είπα, ο κύριος Τιμπορσάνη είναι ο εισηγητής, αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εμείς θα συντάξουμε γνωμοδότηση. Και φέτος, όπως και πέρυσι, η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα εκπονήσει έκθεση με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εντολή ε, και για το φετινό τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό. Πρόκειται για τη θέση μας, τις πρώτες μας αντιδράσεις σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του 2018. θέλουμε μέχρι τις 23 ε, Απριλίου να υποβληθούν, 26 ε, Απριλίου να υποβληθούν οι τροπολογίες στη μία η ώρα, 29, 29 και 30 Μαΐου θα ψηφίσουμε, θα εγκρίνουμε το σχέδιο γνωμοδότησης, ώστε ε, να τη δώσουμε εγκαίρως στην Επιτροπή Προϋπολογισμών που είναι αρμόδια κατ' και θα ψηφίσει 19 με 20 Ιουνίου. Αυτά και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Τίμπορ Σάνι για να μας ε, παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο ε, αυτής της διαδικασίας. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε αυτής εξ αρχής ότι ο ρόλος της γεωργίας, εκτινοτροφίας και ανάπτυξη πέθρου είναι σημαντικό για την υιοθέτηση πολλών ε, στόχων προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτά που αναφέρω στην γνωμοδότησή μου και οι τομεί που αναφέρω θα μπορούσαν να, ε, να διευρυθούν επαόριστον. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ως προς τα αιτήματα του γεωργικού κλάδου για τον προϋπολογισμό του 2018. Στο σχέδιο γνωμοδότησης, που είναι βέβαια ένα τεχνικό έγγραφο, ε, περιλαμβάνω και κάποια νέα σημεία που θα πρέπει να ενισχυθούν, όπως ε, η μνήμα της ρήτρας του ενεργού γεωργού των ε, ομάδων παραγωγών και της καταπολέμησης των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Πιστεύω κράτοντα ότι μπορούμε να βρούμε ευφύης λύσεις και στη γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, γιατί θεωρώ σημαντικό να αναζητήσουμε τέτοιες ευφύης λύσεις, όπως επισημαίνω και στην έκθεση. Πάντως, στην γνωμοδότησή μου χαιρετίζω τα νέα παρατηρητήρια αγοράς και προτείνουμε ε, περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της προσέγγισης και διεύρυνση στις... Περιμένω τις τροπολογίες σας, συνάδελφοι, και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία με τους κοιόδης ηγετές, αλλά και με όλους τους ε, ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Μάλιστα, θα ανταποκριθούν ε, οι ευρωβουλευτές ε, στην πρόσκλησή σας Πρώτα η κυρία Μπεάρτερ. Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Μπέλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Σας ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα πρότασή σας. Εγώ είχα κάποιες παρατηρήσεις και θα ήθελα να τις κάνω αυτής εξ αρχής. Ένας ισχυρός προϋπολογισμός για τη γεωργία. Δεδομένου όμως ότι αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικές ε, προκλήσεις, θα μπορούσαμε ίσως στη γνωμοδότησή σας να προσθέσουμε ότι θέλουμε ένα προπολογισμό που να είναι τουλάχιστον στο ύψος του προηγούμενου έτους. Δεύτερο που θα ήθελα να πω αφορά την απλοποίηση. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να επιμείνουμε ότι η απλοποίηση των κανόνων είναι κάτι το απαραίτητο. Τρίτο, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αναφερθήκατε στις οργανώσεις παραγωγών στην παρουσίασή σας. Οι κανόνες δεν είναι πάντα βέβαια πάρα πολύ σαφείς και αυτό φοβίζει τους αγρότες οι οποίοι θέλουν πολλές φορές ε, μέσω αυτών των ενώσεων να κατανοήσουν καλύτερα το τι ε, ακριβώς προβλέπουν οι κανονισμοί. Τους θεωρούν εξαιρετικά περίπλοκους. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι σαφές για μας, γιατί η χρήση αυτών των ε, ε, ποσών προϋποθέτει την κατανόηση από μέρους των παραγωγών και των γεωργών των κανόνων. Ο κύριος Ανδρέα, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Τίμπορ για την δουλειά του και να επιμείνω σε ένα σημείο. Αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ για το 2018 που αφορούν τις σημερινές κρίσεις δημόσιας υγείας, υγείας των ζώων και των φυτών. Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την γρήπη των πουλερικών σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από αυτή που μας έπληξε τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε στην καρδιά αυτής της κρίσης και την ίδια ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και η πανόλη των χείρων. Εγώ πιστεύω και επιμένω ότι αυτό το ποσό σίγουρα δεν αρκεί για το 2018. Και θα ήθελα να πάρω το λόγο επίσης για να σας πω ότι χρειάζεται λόγω μια πιλωτική δράση για, την, ε, για τον τομέα του ίνου και της αμπελουργίας. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αμπέλια. Κάθε χρόνο 8 με 10% της παραγωγικότητας αυτού του τομέα μειώνεται. Και δεν είναι ένα μικρό πρόβλημα αυτό για τους ε, αβελουργούς και τους συνοπαρακογούς. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, θερμά τον εισηγητή και για την πρόταση που κατά τη εκείνος και για όλες τις άλλες προτάσεις. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα θέματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ε, να διατηρήσουμε τον προπολογισμό που έχουμε καταρτήσει για τη γεωργία. Πρέπει να πολεμήσουμε γι' αυτό. Εγώ δεν θέλω να υπάρχουν συνεχώς μεταφορές σε άλλους τομείς. Αυτό που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ότι τα κονδύλια που αφορούν στην κρίση, κατά κανόνα, αυτά εκταμιεύονται κάθε χρόνο για περιπτώσεις, για προβλήματα που δημιουργούνται ακριβώς λόγω κρίσης. Ε, δεν ξέρω, αυτό είναι αυτό που εννοούμε στο σημείο υπαριθμών 3. Κάτι άλλο που θέλω να συζητήσουμε είναι οργανώσεις παραγωγών. Γιατί ε, βασικά δεν είναι δύσκολο να συσταθεί μια οργάνωση παραγωγών. Ε, όταν πρόκειται για να ε, χρησιμοποιηθούν κονδύλια για τη δημιουργία ενώσεων παραγωγών μέσω του leader και άλλων προγραμμάτων, αυτό μπορεί να γίνει. Εκείνο όμω που θέλω να μου εξηγήσει τελικά, είναι αυτό που λέτε ευφυεί λύσει. Ευφυεί λύσει τι είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω καλά. Και η σημασία των πιλωτικών σχεδίων. Ε, από τη δική μου εμπειρία ε, μπορώ να σας πω ότι τα πιλωτικά προγράμματα δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν μόνο για δύο χρόνια για να δημιουργήσουν κάποιες θέσεις απασχόλησης και μετά ε, εξαφανίζονται. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή ότι τα πιλωτικά προγράμματα είναι και αποτελεσματικά. Ίσως θα πρέπει να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες από αυτού. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και επίσης ε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κυρίως ε, διότι η γνωμοδότησή του είναι ευσύνοπτη, είναι αποτελεσματική. Πράγματι, φίλε, έμεινε στην ουσία του θέματος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ χαιρετίζω τα παρατηρητήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 και στο άρθρο 9 ε, πράγματι αυτά που αναφέρονται είναι θετικά, δηλαδή το να μπορούμε να ε, προβλέψουμε κάποιες καταστροφές και να προσφέρουμε κάποια προστασία. Αυτή τη στιγμή προβλέπουν 20 εκατομμύρια για αυτόν τον σκοπό. Αν δεν φτάσουν θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσό. Όσον αφορά τώρα στις αντίστοιχες και οδών εισηγητών, ε, σχεδόν συντονιστών. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνουν αυτές. Έχω τρει-τέσσερι ερωτήσεις να κάνω. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείται στο άρθρο 2, εκεί που γίνεται λόγος για το υπάρχον περιθώριο της γεωργίας, αυτό να είναι συγκεκριμένα συνδεδεμένο με ένα στόχο. Τι εννοείται συνδεδεμένο με ένα στόχο, θέλω να το καταλάβω αυτό. Με τα άρθρο 3 πρόκειται για τη ρήτρα των ενεργών ε, ιδιοκτητών γεωργικών μονάδων. Θα θυμάστε ότι στην τελευταία μεταρρύθμιση Διαφωνήσαμε διαμακρών από αυτού, διότι τότε ο Επίτροπος Τσόλος ήθελε να δημιουργήσει έναν νέο ορισμό. Μετά όμως αυτός δεν μπορούσε να μεταφραστεί. Ε, χαίρομαι που το συζητήσαμε ή και θα το συζητήσουμε το τι ακριβώς είναι αυτό το ενεργός ιδιοκτήτης. Ε, κυρία Μίλλουρ είπε στο άρθρο 6 εκεί που γίνεται λόγος για ευφυείς λύσεις. Εγώ θα ήθελα να μην μιλάτε μόνο για ευφυείς, να μιλάτε για ευφυείς και καινοτόμες λύσεις για να ικανοποιηθώ. Και επίση ε, και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι είπαν ότι ο προπολογισμό ε, τη Γεωργία θα πρέπει να παραμείνει σταθερό Λόγω του ότι θα έχουμε και το Brexit, ε, πρέπει να πούμε ότι ε, κατά τη διάρκεια του διαζυγίου η Βρετανία εξακολουθεί να έχει δικαιώματα και υποχρώσεις. Ε, ως εκ τούτου, μέχρι το τέλος ε, της θητείας θα πρέπει, μάλλον μέχρι να αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να διαθέτει και αυτή τα απαραίτητα κονδύλια στον ε, ενωσιακό προεπλογισμό. Βλέπω ότι νεύεται καταφατικά και χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, Μάλιστα. Ο κύριος Τιμπόρ φαντάζομαι πήρε παράδειγμα από τη, από δική σου γνωμοδότηση που επίσης ήταν πολύ συγκεκριμένη και άρτη. Ο κύριος Νίκολσον, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ακούω ε, αυτό το εφής και να είστε εφής και να είστε έξυπνος, εύκολο είναι να είναι κανείς εφής στις Βρυξέλλες, αλλά τα έξυπνα υποτίθεται εφή, αυτά τα προγράμματα πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα αγρόκτημα. Και εκεί είναι που κολλάνε εξαιτία της γραφειοκρατίας και των ε, διοικητικών διατυπώσεων που παρεμποδίζουν τους γεωργού στο έργο του. Επίση, όλοι γνωρίζουμε ότι με την κρίση στο γαλακτοκομικό κλάδο και όλε τι κρίσει που βιώσαμε, χρειαζόμαστε παροχή πληροφοριών και ταχύτερα από τα κράτη-μέλη, αλλά αξιόπιστων πληροφοριών. Και αν συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο, και αν θα έχουμε και θα ιδρύσουμε νέους φορείς, θα πρέπει πρώτα να διαλύσουμε τους παλιούς φορείς. Έτσι θα μειώσουμε και το κόστος. Θέλω λιγότερη επικάλυψη, γιατί αυτό είναι που κάνουμε. Πολλαπλασιάζουμε φορείς ε, με αποτέλεσμα να ενισχύουμε την επικάλυψη. Έχουμε όλο, περισσότερου όλο περισσότερους νέους φορείς ε, που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους γιατί οι παλιοί εξακολουθούν να υπάρχουν, δεν έχουν αργηθεί. Οπότε αυξάνεται η επικάλυψη. Θέλουμε να μειώσουμε την επικάλυψη. Το είδαμε και προηγουμένως στη συζήτηση για τις κλιματικές αλλαγές. Είναι τρομακτικά αυτά που μας περιμένουν ή που δεν μας περιμένουν. Θα εξαρτηθεί. Πάντως έχουμε καθήκον να αφήσουμε το περιβάλλον ε, στις επερχόμενες γενιές, σε, σε επερχόμενες γενιές τουλάχιστον σε, στην ίδια κατάσταση, αν όχι σε καλύτερη από αυτή που την πήραμε εμείς. Και θα πρέπει να ξοδέψουμε και περισσότερα κονδύλια εκεί που χρειάζεται. Γιατί πολλέ φορέ ακούμε για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος μπορεί να ξοδέψει χρήματα σε πολλούς τομείς, σε πολλά θέματα, αλλά αν έχει και κάποιο κέρδο. γιατί αν δεν του μείνει κανένα κέρδο και δεν μπορεί να ε, επιβιώσει, πώς θα αναλάβει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Αν ένας έχει μια γεωργική επιχείρηση και δεν έχει αρκετά χρήματα να αγοράσει φαγητό για την οικογένειά του, να κάνει το καθήκον του, τότε τι θα θυσιάσει πρώτα. Θα θυσιάσει αυτές τις ώρες ε, ευφυείς, ε, μεγαλεπίβολες και φιλόδοξες ιδέες. Συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, να εξασφαλίσουμε κονδύλια ε, για να προσ... Θα προσφέρουμε στους γεωργούς. Αλλιώς δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υλοποιήσουν όλες αυτές τις δράσεις. Ε, μας προσγείωσε ο κύριος Νίκολσον στην πραγματικότητα με αυτά που είπε. Για να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε την κοινή γεωρική πολιτική θα πρέπει να έχει κανείς ε, ένα επίπεδο νοημοσύνης. Και αυτό πραγματικά το έχουν οι γεωργοί και το κάνουν πολύ καλά. Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη ότι σε ό,τι αφορά την νοημοσύνη και την καινοτομία, ο Γιώργος θα καταφέρει μια χαρά και μερικές φορές δεν χρειάζεται την έμπνευση και τον ίστρο των Βρυξελών. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο ή την εκπρόσωπο της ε, ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σχολιάσει. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την σοφή και σύντομη έκθεση και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική και σαφής. Αυτό είναι το μόνιμο δίλημα, να σχολιάζουμε πράγματα που δεν έχουμε δει ακόμη. Ακόμη δεν έχει υποβληθεί το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018, οπότε και εγώ έχω το δίλημα πώς να σχολιάσω τα σχόλιά σας για κάτι που δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί. Ελπίζουμε ο προπολογισμό, το σχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίζει αρκετή χρηματοδότηση για την εφαρμογή τη κοινή ζωρική πολιτική, όπω είχε συμφωνηθεί στην ε, μεταρρύθμιση του 2013. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να ξαναδιαμορφώνουμε την κοινή γεωργική πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για να συμπεριλάβουμε και νέες πρωτοβουλίες που δεν είχαν συμφωνηθεί στη μεταρρύθμιση του 2013. Βέβαια, όλη η προσπάθεια του Επιτρόπου Χόγκαν και των υπολείπων επιτρόπων ε, για την απλούστευση θα φέρουν ένα φρέσκο αέρα στην Επιτροπή, μια νέα πνοή ανέμου αλλά μην ξεχνάτε ότι μας ε, περιορίζει το πλαίσιο μεταρρύθμισης του 2013. Πάντως, το σχέδιο προϋπολογισμού που θα σας ε, υποβάλουμε το Μάιο θα προβλέπει αρκετή χρηματοδότηση για τις άμεσες ενισχύσεις. Αυτές οι άμεσες ε, πληρωμές, άμεσες ενισχύσεις θα εφαρμοστούν για τρίτη συνέχεια χρονιά και ευελπιστούμε ότι με την εμπειρία που αποκομίσαμε από τα δύο προηγούμενα χρόνια εφαρμογής, το 2016 και το 2017, η εφαρμογή επιτόπου των άμεσων ενισχύσεων θα είναι πιο βελτιωμένη. Αυτό φαίνεται και στις, στα αιτήματά μας για τον προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες της αγοράς, θα διαπιστώσετε μία μικρή μείωση σε σχέση με το 2016 και 2017. Τα πακέτο των 500 εκατομμυρίων που υιοθετήσαμε το 2016 και 2017 δεν θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό του 2018 πια. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει το αίτημα για συνεχή μέτρα για τα οποροκυπευτικά ε, παρά τις μειωμένες ανάγκες, γιατί πρόκειται για την τέταρτη πια χρονιά εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά τις επιζωτίες, τα κρούσματα επιζωτιών και άλλες πιθανές κρίσεις αγοράς, ε, θα συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, στις αγορές. Σε περίπτωση που χρειαστούν δράσεις, έχουμε και τη δυνατότητα του, της διορθωτικής επιστολής για τον προϋπολογισμό που θα υποβάλουμε το φθινόπωρο. Θα έχουμε και εκεί την ευκαιρία, αν χρειαστεί, να ε, προτείνουμε αυξήσει κάποιων κονδύλιων. Επαναλαμβάνω, αν παραστεί ανάγκη. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα, θα αυξηθούν οι ανάγκες πληρωμών σε σχέση με το 2016 και 2017, μια και τα προγράμματα έχουν ε, μπει σε κανονική ταχύτητα εφαρμογής και προχωρούν καλά στην εφαρμογή τους. Το θα, έχει κλείσει το, θα έχουν κλείσει τα προγράμματα και από την παλιά περίοδο, οπότε από αυτό θα προκύψουν νέε ανάγκε. Και σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, τα πιλωτικά σχέδια, όπω πάντα, μα ε, ενδιαφέρουν και περιμένουμε τι προτάσει σα για τα πιλωτικά σχέδια. Και πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο προϋπολογισμού θα τύχει της υποστήριξης της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οπότε φαίνεται ότι έχετε παρόλα αυτά καλύτερη ενημέρωση για τον προϋπολογισμό. Αυτό φάνηκε από τα σχόλια που κάνατε. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την πρόταση του προϋπολογισμού. Όπως ξέρετε, οι αγορές επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες ή από τις καιρικέ συνθήκες και από τις κρίσεις που ενσκύπτουν και εξαρτάται από ποια περίοδο του έτους εμφανίζονται οι κρίσεις. Ε, ανάλογα τις αντιμετωπίζουμε και με τα διάφορα μέτρα. Αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο και πάλι στον εισηγητή, στον συντάκτη γνωμοδότησης, για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Σάνι, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις σας. Για λόγους που αφορούν ρυθμιστικά θέματα, είναι τεχνικά και όχι τόσο πολιτικά τα θέματα. Οι, ερω... οι προτάσεις μας πρέπει να είναι προτάσεις που να καλύπτουν όλο το φάσμα και βεβαίως αυτό μπορεί να σας φανεί πρακτικό πρόβλημα, αλλά δεν το ξεπεράσαμε και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αν θέλετε, οι προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες ε, προετοιμάστηκαν εκ παραλίλου με τις δικές μας προτάσεις και προτιμήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σίγουρα θα το επεξεργαστούμε εκ νέου. Και φανταζόμαστε, ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της αυτές τις προτάσεις. Τώρα, δύο λόγια σε σχέση με αυτά που άκουσα από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Εννοείται ότι εγώ είμαι ανοιχτός στις δικές σας απόψεις και προτάσεις. Εδώ εκφράζουμε την άποψη του Κοινοβουλίου. Μου λέτε για την απλοποίηση, το καταλαβαίνω. Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα που αφορούν την υγεία. Θέλουμε να αντικατοπτρίσουμε και τις αδυναμίες του συστήματος. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Το θέμα των ορισμών, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθοριστικό. Ελπίζω να φτάσουμε κάποια μέρα σε καθαρούς ορισμούς. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το μέχρι τώρα ισχύον σύστημα. Χρειάζονται βελτιώσεις στους ορισμούς, εννοείται. Και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Και η Επιτροπή πιστεύει ότι τα πιλωτικά προγράμματα έχουν καθοριστική σημασία. Αυτά τουλάχιστον που θα συνεχιστούν. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα και έχει αποτελέσματα, και όσον αφορά τα έξυπνα προγράμματα, υπήρξαν σχόλια για αυτό το θέμα. Τι ακριβώς είναι αυτό το έξυπνο όταν αναφερόμαστε στην ε, Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους. Καταλαβαίνω ότι μετά από αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε, το πιο σημαντικό είναι η αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν σε αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Σάνι. Επαναλαμβάνω τις τροπολογίες να τις στείλετε μέχρι τις 26 Απριλίου, μία το μεσημέρι, στο γραφείο του συντάκτη της Γρομοδότησης. Σας ευχαριστώ θερμά. Μπορεί να μην έρθετε όλοι αύριο. Όποιοι είναι σήμερα αλλά θα απουσιάζουν αύριο, να τους ευχηθώ από τώρα χρόνια πολλά για το Πάσχα. Οι υπόλοιποι θα συνεδριάσουμε αύριο 9 το πρωί με 12.30 και 3 το απόγευμα. Ελπίζω να τελειώσουμε νωρίτερα το απόγευμα. Αυτό θα προσπαθήσω πάντως. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.